Uh, good morning everyone. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ω συνήθω, το πρώτο σημείο είναι η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ε, η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη ε, άλλη τη Δευτέρα. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρείται ε, χωρί αλλαγέ ε, εγκεκριμένη. Καταρχήν, να σα ενημερώσω για τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Καταρχήν για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ο πέμπτος τριμερής διάλογος για, το, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος, τέταρτη φάση. Εξετάζονται διάφορες πτυχές του θέματος, όπως την ενημέρωση της οδηγίας για την ρήπαση από τα οχήματα και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, την προστασία κατά της διαρροής του άνθρακα και ούτω καθεξής. Είχαμε εκτενείς συζητήσει ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων ως προς το πακέτο με ε, διάφορες συμβαστικές προτάσεις και παρά τη, τον επικοδομητικό διάλογο και τις έντονες προσπάθειες των θεσμικών οργάνων να, να καταλήξουν συμφωνία, τελικά αποτελματώθηκαν οι διαπραγματεύσει ό,τι αφορά τη συμπερίληψη ε, των προδιαγραφών για τις επιδόσεις ως προς τις εκπομπές. Δεύτερον, ε, σύστημα εμπορίας εκπομπών για την ε, αεροπορία. Χθες έγινε τελευταίος τριμερής διάλογος για την εμπορία εκπομπών στην αεροπορία. Συμφωνήσαμε σε πολλά σημαντικά θέματα όπως είναι ε, η τρέχουσα εξαίρεση, να παραταθεί μέχρι την 21 η Δεκεμβρίου ε, το 2023. Επίσης, ε, προσδιορίστηκε το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες για την αναθεώρηση. Το 15% πληστηριασμού των δικαιωμάτων θα περιληφθεί στη μεταρρύθμιση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδήλωσε την πρόταση ε, την πρόθεση να προτείνει αύξηση του ποσοστού αυτού του 15% και η, ασφαλιστική, δικλίδα για την προστασία της ακεραιότητας ε, του ETS συμπεριληφθήκε με την τελευταία, συμπερίληψη του τελευταίου πρόταση του Συμβουλίου για τις ε, ε διατάξεις GATT. Οπότε ε, αναφέρθηκε ανάγκη η ΚΑΟ να δράσει με απόλυτη διαφάνεια ε, και να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, ε, η, η επιλογή για τις ε, κατεξοδότητες πράξεις για τα θέματα MRV θα αποφασιστούν στην τέταρτη φάση, στον επόμενο τριμερή διάλογο, γιατί αυτός, αυτό το θέμα αποτελεί τμήμα της γενικής αξιολόγησης του ETS. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις ως προς τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Μερικές ανακοινώσεις τώρα. Εξής μία. Μετά την απόφαση της Ολομέλειας να παραπέμψω το θέμα του επιμερισμού των προσπαθειών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και με βάση το άρθρο 69F η διαπραγματευτική ομάδα με ε, την υποφαινομένη ως πρόεδρο και ε, παρουσία του εισηγητού Γκριμπάλτη και των σχεδόν εισηγητών έχετε λάβει όλοι ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ε, τα έγγραφα της συνεδρίας και έχουμε και διερμηνία σε 20 γλώσσες. Πρώτο θέμα της της διάταξης, υποβολή αντιρρήσεων. Σε ό,τι αφορά ε, την την εκτελεστική πράξη για την παράταση της προθεσμίας για την έγκριση του, της γλυφοσάτης. Ε, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη το υπόβαθρο της πρότασης αυτής. Πρόκειται για διαδικασία αντίρρησης. Ίσως όμως καλύτερα να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές για να μας ενημερώσουν. Πρώτα τον κύριο Παύλ Πότς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα τσεχικά, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, την κυρία Κόνετσνα, τον κύριο Εκχόουτ, τον κύριο Πεντοτσίνη, την κυρία Εύη και τον κύριο Γιάκ και να επισημάνω ότι, όπως είπε η Πρόεδρος, υποβάλαμε με βάση το άρθρο 106 ε, ένσταση αντίρρηση για, τον, ε, ε, για την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τον κανονισμό 1107 του 2009 σε ό,τι αφορά τη θέση σε εμπορία στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γλυφοσάτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε παράταση της άδειας για την γλυφοσάτη για μία ακόμη δεκαετία, παρόλο που η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί από τις 20 Ιουνίου, μέχρι στιγμής δεν έχουμε συγκεντρώσει την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία. Κάτι που δεν εκπλήσει διόλου, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο παρελθόν είχε προτείνει παράταση κατά μία ενιαετία της άδειας για την γλυφοσάτη, παρόλο που η Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων είπαν ότι είναι υπέρ της παράτασης της άδεια, φαίνεται ότι και η ΕΦΣΑ και η άλλη εταιρεία αγνοούν τις αντενδείξεις για τη χρήση του προϊόντος αυτού. Γιατί αναφέρθηκε ότι δεν έχει καρκινογόνα αποτελέσματα γλυφοσάτη λόγω της περιορισμένης χρήσης της, αλλά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου εκρεμεί δίκη α, με, μετά από μηνύσεις που έγιναν από ασθενείς με λέφωμα Χότσκινγκ. Ε, επίσης διέρευσαν κάποια έγγραφα από τη Μονσάντο που δημιουργούν πολλές αμφιβολίες ε, και επιφυλάξεις για κάποιες μελέτες που είχε ε, αναθέσει η ίδια η Μονσάντο ε, και αποτέλεσαν και τη βάση για τις μεταγενέστερες μελέτες της ΕΦΣΑ και του ΕΚΑ. Χρειαζόμαστε σαφή και αξιόπιστα στοιχεία, αμερόληπτα. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 1-3 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν κατάργηση, απαγόρευση της χρήσης γλυφοσάτης. Για να μην μιλήσουμε κάποιους ισχυρισμού για ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ε, κάποιες μελέτες του 2016 μιλούν για αύξηση του κινδύνου καρκίνου του δέρματος, μελανόματος ή αύξηση της χρήσης ε, με κοιτοκτόνων και ζυζανιοκτόνων σε συνδυασμό με την ε, παρατεταμένη έκθεση στην ηλιοφάνεια. Επίσης, άλλη μεταανάλυση του 2016 μιλά για έκθεση στη γλυφοσάτη που, που προκαλεί αύξηση της, των πιθανότητων να προσβληθεί κανείς από λεύχομα Χότσκινς ή λευχαιμία. Επίσης, κάποια εμπορικά προϊόντα, όπως το Δεκάμπα, περιέχουν γλυφοσάτη. Και τέτοια προϊόντα αλλάζουν την ε, δεκτικότητα του σώματος ε, ε, στα αντιβιωτικά και άρα κάνουν το σώμα πιο ευάλωτο απέναντι στα βακτηρίδια. Η γλυφοσάτη σε μικρές δόσεις χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού, κάτι που μπορεί να οξύνει το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής. Αυτό όμως δεν αναφέρθηκε διόλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη έχουμε και αμεταλφοσφορικό και μεταφοσφωνικό οξύ που μπορεί να βλάψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο σώμα του ανθρώπου. Ούτε αυτά τα στοιχεία έλαβε υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντα την παράταση της άδειας για τη γλυφοσάτη. Ο κανονισμός 1107 του 2009 προβλέπει ότι τα μέτρα του θα πρέπει να εδράζονται στην αρχή της προφύλαξης και στην αποτροπή οποιονδήποτε αρνητικών αποτελεσμάτων στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία των αντιρρήσεων, των εστάσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη τα σχόλιά μας. Ήδη το 2016 ζητήσαμε άμεση απαγόρευση της χρήσης γλυφοσάτης κοντά στα δημόσια πάρκα ε, και ζητήσαμε να απαγορευτεί η γλυφοσάτη ε, σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται η αρχή της ολοκληρωμένης προστασίας των φυτών. Επίσης, προτείναμε σταδιακή μείωση ε, της χρήσης της την επόμενη τριετία μέχρι την κατάργηση και δώσαμε συγκεκριμένες ε, ε, προτάσεις για πιθανή συμβαστική λύση. Για παράδειγμα, μεταβατική περίοδο για τους γεωργούς και πρώτα απ' όλα ανεξάρτητη και το τονίζω ανεξάρτητη αμερόληπτη μελέτη για τη γλυφοσάτη, κάτι που δεν συνέβη μέχρι στιγμής. Η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ χρησιμοποίησαν τις ίδιες μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια την Μονσάντο, την εταιρεία που παράγει τη γλυφοσάτη και άλλους εμπορικούς εταίρους της. Χρειαζόμαστε φυσικά τους οργανισμούς ε, όπως είναι ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων και η ΕΚΑ, αλλά θα πρέπει να ε, εκτελούν σωστά το έργο τους. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι με την ε, πρότασή μου, γιατί μερικές χώρες θέλουν παράταση όχι μόνο για άλλη δεκαετία, αλλά επάπειρον και χωρίς καμία, κανένα περιορισμό για τα ζυζανιοκτώνα. Μάλιστα, μερικές φορές χρησιμοποιείται ως αποξηρατική ουσία πριν την εσοδεία, κάτι που είναι ό,τι χειρότερο. Εμείς απο... απορρίψαμε τέτοια χρήση για την γλυφοσάτη και τελικά το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν περιλήφθηκε τελικά στον κανονισμό. Πάντως, με βάση τη στάση πολλών κρατών μελών και αν δεν ευοδοθεί η διαδικασία έσταση, θα πρέπει να επανέλθουμε ε, ξανακαταθέτοντας την. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, θεωρεί έγκυρες αυτές τις ενστάσεις μας, αλλά παρακαλώ η Γενική Διεύθυνση Υγείας ε, να λάβει υπόψη τις πληροφορίες που έχουμε και που λέει ότι η γεωργοί που χρησιμοποιούν γλυφοσάτη θα προσφύγουν στο δικαστήριο κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από φόβο να αποφύγει τέτοια δίκη πρότεινε παράταση της άδεια γλυφοσάτη για μια δεκαετία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόκειται στον έμεσο εκβιασμό των παραγωγών γλυφοσάτη. Ελπίζω να συμφωνήσετε με τη διαδικασία αντιρρήσεων για την απόρριψη τη. σα. ευχαριστώ. λεπτά, αλλά έχουμε περιορισμένο χρονικό διάστημα, γι' αυτό λοιπόν ε, Προσθέθηκε αυτό το θέμα στην ημερήσια διατάξη σήμερα. Ω προσθήκη λοιπόν έχουμε ψηφοφορίες. Θα ήθελα σας παρακαλώ να δείξετε αυτοπιθαρχία. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Μην επαναλαμβάνετε όμως τα επιχειρήματα που έχουμε ήδη ακούσει. Να είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε και κατάλογο μελητών. Δεν θέλω να διακόπτω κανέναν. Η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την έγκριση της γλυφοσάτης είναι προηγουμένου. πραγματικά αηδία. Ε, Νιώθω. Και τι να σας πω, ε, ε, αηδιασμένη ήμουν πριν από έξι μήνες. Τώρα πλέον έχω περάσει στο επόμενο επίπεδο. Η ακαδημαϊκοί κύκλοι και επιστήμονες εξακολουθούν να υποδεικνύουν τις επιζήμιες συνέπειες της γλυφοσάτης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να κοφεύει και θέλει να δώσει έγκριση στη γλυφοσάτη με οποιοδήποτε τμήμα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Εμείς δε έχουμε δει διάφορα σκάνδαλα σε ό,τι αφορά τη Μοντσάντο, σε ό,τι αφορά την επιρροή που έχουν στις επιστημονικές ε, μελέτες και έρευνες. Και έχουμε ήδη αναφέρει Τη επικοινωνία που έχουν διαρρεύσει σε ό,τι αφορά την εταιρεία αυτή και έχουμε δει ότι έχει δώσει και αναθέσει τη διεξαγωγή μελετών, τι οποίε μετά παρουσιάζει ω ανεξαρτητε Επί 17 και πλέον έτη, η εταιρεία αυτή γνωρίζει ότι ενδεχομένω δεν είναι επιζήμια αυτή η ουσία και παρόλα αυτά δεν έχει κάνει τίποτα. Παρά λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα, παρά όλα αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει. Προσπαθεί λοιπόν να αποφύγει πάση θυσία οποιοδήποτε δημοκρατικό έλεγχο και η εφαρμοστική πράξη μας κατατέθηκε με καθυστέρηση χωρίς να έχουμε χρόνο ουσιαστικά να προετοιμάσουμε τις αντιρρήσεις μας. Χρησιμοποιεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την διαδικασία προσπαθώντας να αποφύγει το δημοκρατικό έλεγχο και γι' αυτό λοιπόν υπέβαλαν την πρόταση τόσο καθυστερημένα. Δεν θέλουν πολύ απλά να ακούσουν οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, οποιαδήποτε αντίρρηση και εμείς συνεχίζουμε να προβάλλουμε αντιρρήσει. Η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε εσφαλμένα, αναλυθή επιστημονικά στοιχεία, προσαρμοσμένα στα συμφέροντα του κλάδου. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράσει τώρα, εδώ και τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αγνοεί, αγνοεί παντελώ ε, τι πρωτοβουλίε των πολιτών, αλλά θα αναγκαστεί να ακούσει την φωνή ενός εκατομμυρίου και πλέον ε, Ευρωπαίων πολιτών που έχουν προσυπογράψει την ε, αίτηση για την απαγόρευση της γλυφωσάτης. Πριν από κάποιες εβδομάδες, ε, πριν από κάποιους μήνες, ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα πιστήρια της Μονσάντο, τα τεκμήρια της Μονσάντο πιο ενδελεχώς. Αρνήθηκε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει ότι καταφανώς άγνοη και περίφρονε την αλήθεια. Και θέλω λοιπόν να ερθώσουμε το αίσθημά μας. Επόμενος μελητή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έκχαουτα, να προσθέσω στα επιχειρήματα τα οποία μόλι ακούσαμε εδώ το εξή. Νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ασφαλώ γίνεται μια τεράστια συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα για τι τις ιδιότητε τη της Είναι όμω επίση σημαντικό ότι γνωρίζουμε ότι η γλυφωσάτη πραγματικά σκοτώνει την περιβαλλοντική διάσταση και ζωή. Το θέμα δηλαδή δεν είναι ότι η γλυφοσάτη έχει πατέντα ως ε, αντιβιωτικό. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο και στο ΕΚΑ. E Επίσης η ΕΚΑ e καταλήγει στο πόρισμα ότι είναι τοξική η γλυφοσάτη για το υδρόβιο περιβάλλον σε μεγάλο χρονικό διάστημα και ξέρω ότι οι συζήτησεις συχνά εστιάζονται στην κατά πόσο είναι καρκινογόνος ουσία ή όχι. Αυτό είναι αφιλεγόμενο. Υπάρχουν πολλές ε, αμφιβολίες, αλλά ισχύει και η αρχή της πρόληψης, αλλά κοιτώντα την επίδραση στα ζώα, στην Πανίδα και στη Χλωρίδα, τη Θαλάσσια και τη Χερσαία, η Κίδιο και η ΕΦΣΑ, είναι καταφανώς ε, και κατηγορηματικά άμα, σίγουρες ότι πρόκειται για μόλυνση και χρειάζεται χρόνος προσαρμογής και γι' αυτό λοιπόν στο ψήφισμα αυτό διευκρινίζουμε ότι μέχρι το τέλη του χρόνου μπορούμε να το να χρησιμοποιούμε και συχνά λέμε ότι χρειάζεται μια τριετής μεταβατική περίοδο για να υπάρχει σταδιακή κατάργηση στην εμπορική χρήση παράλληλα με την γεωργική χρήση. Ξέρουμε λοιπόν ότι τους δίνουμε χρόνο. Συνολικά, αυτά που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα έχουν πολύ πιο πολύ νόημα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δεκαετή ανανέωση της έγκρισης. Τελευταίο στοιχείο, κυρία Πρόεδρε, και αυτό το απευθύνω σε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν έλαβε κατευθείαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μην μας πείτε ότι α, μπορούσατε να κοιτάξετε στην ιστοσελίδα. Ξέρουμε ότι το στείλατε στο Συμβούλιο προς και δεν απεστάλλει παράλληλα και προς το, προς το Κοινοβούλιο. Αυτό η Επιτροπή να μας το εξηγήσει. Γιατί αυτό προκαλεί τη μεγάλη χρονική πίεση που έχουμε αυτή τη, στιγμή και όλους μας ενοχλεί και εσάς σαν πρόεδρο προφανώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Έικαουτ, ο κύριο Σπεντιτσίνη, από το EFD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με αυτά που είπε ο συνάδελφο Αϊκάουτ έστω και αν από τη δικιά μας άποψη ε, εμείς θα είμαστε πάντα αντίθετοι σε οποιαδήποτε είδους ανανέωση της ε, αδειοδότησης. Ωραία, πρέπει να συζητήσουμε για μια μεταβατική φάση. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα πρέπει, είναι απαραίτητη μεν, αλλά θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη. Παραπέρα εμείς δεν μπορούμε να πάμε, όχι μόνο για ε, λόγω όλων αυτών τα, ε, που αναφέρθηκαν ήδη σχετικά με το θέμα αυτό, αυτό, δηλαδή την αδυναμία ε, των οργάνων απέναντι σε μια ισχυρή πολυεθνική και για την ε, διεθνή μας θέση, αλλά ε, κατέδειξε επίσης ε, την ανεπάρκεια των συστημάτων μας απέναντι στη διαφάνεια, απέναντι στη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τα επιστημονικά τεκμήρια. Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι από μια περιοχή την οποία επισκέφθηκα και πρόσφατα και διαπιστώνει κανείς εκεί ε, ότι η γλυφοσάτη η οποία χρησιμοποιείται δίνει την δυνατότητα σε βόρειες ε, περιοχές ε, να καλλιεργήσουν σκληρό σύτο με δυνατότητες και με τρόπους τέτοιους όμως που καταστρέφουν τις ντόπιε καλλιέργειες. Είδαμε λοιπόν ότι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ε, παρήγαγαν σκληρό σύτο ε, για την εσωτερική παραγωγή ζυμαρικών αλλά και ε, για, εξαγωγές είτε έκλεισαν είτε χρειάστηκε να πάνε προς το βορρά και φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου αναγκαστήκαμε να κάνουμε εισαγωγή σύτου από τον Καναδά. Δεν είναι δυνατόν ούτε οικονομικά ούτε με άλλο τρόπο μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη χωρίς να επαναλάβω οτιδήποτε είπαν προηγούμενοι ε, συνάδελφοι γιατί και εγώ είμαι, ε, έχω προσυπογράψει αυτό το θέμα ε, για την γλυφοσάτη ε, σε μία ακόμα, σε ένα ακόμα κείμενο, σε ένα ακόμα ψήφισμα από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μας. Είχαμε μάλιστα και μία ακρόαση στην Επιτροπή Γεωργίας όπου επί τρεις ώρες Ακούσαμε την επιχειρηματολογία των διαφόρων οργανισμών που όμως δεν μας έμαθαν τίποτα καινούριο. Επί τρεις ε, ώρες ε, ε, είδαμε την, τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων και την ΕΚΑ που μας είπαν τα δικά τους επιχειρήματα, οι υπόλοιποι είπαν τα δικά τους. Δεν φτάσαμε όμως πουθενά. Θα δούμε εάν η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα ψηφίσει ή όχι. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος του έτους. Περιμένουμε ε, να δούμε τι θα γίνει και με το ψήφισμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί εδώ προτείνουμε ένα πολύ λογικό, ε, ε, κάνουμε μια πολύ λογική πρόταση, προτείνουμε ένα πάρα πολύ λογικό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά το phasing out, την σταδιακή απαγόρευση της ουσίας αυτής. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε τις προτάσεις ανανέωσης της Κομισιόν, γιατί εδώ μας λένε συνέχεια «Μα εσείς ε, δεν έχετε δικαίωμα να παρέμβετε, δεν έχετε δυνατότητες». Ε, στο σημείο 1 του ψηφίσματός μας αναφέρουμε σαφώς ότι ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης. Μα αυτό δεν είναι και τόσο ριζοσπαστικό γιατί μας κατηγορούν συνέχεια ότι είμαστε ακραίοι. Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε τον, λόγο, τον, τον τρόπο και τον χρόνο στην βιομηχανία να βρει νέα νέες διαδικασίες. Ε, βεβαίως εμείς ε, ξέρουμε πολύ καλά την κατάσταση, ε, ξέρουμε και ερχόμαστε σε επαφή και με γεωργούς που μας λένε καμιά φορά τι θέλετε να βγούμε με τη φαλτσέτα να κόβουμε τα ζυζάνια στα χωράφια μας. Όχι δεν θέλουμε αυτό και είναι σαφές. Ε, ξέρουμε ποιες είναι οι χώρες, ε, η Γαλλία και η Ιταλία, που από τώρα έχουν ε, πει ότι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα καταψηφίσουν, ελπίζω να υπάρξουν και άλλες. Στο σημείο 7 είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε και τα μέσα και τους σπόρους που είναι απαραίτητοι, έτσι ώστε και η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ να μπορέσουν να κάνουν μια πραγματικά ανεξάρτητη μελέτη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ ως ε, σκιώδης. Έχω μονάχα την κυρία Ντελαέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν θέλω να επιμηκύνω τη συζήτηση. Υπάρχουν πάντων πάντως κάποια ενδιαφέροντα ε, ζητήματα σε σχέση με αυτήν την ε, ένσταση ε, γιατί προσωμιάζει με αυτό που ψηφίσαμε πριν από 18 μήνες περίπου. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει στην ένσταση αυτή, το γεγονός ναι, ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Ναι, το κάναμε αυτό πριν από 18 μήνες και υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δύο επιλογές, ανανέωση ή απόσυρση. Και, θεω... και ε, θα το συζητήσουμε βεβαίως, ε, το phasing out σε τρία χρόνια δεν έχει και μεγάλη έννοια, γιατί είτε πρέπει να ανανεώσουμε, είτε πρέπει να αποσύρουμε. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει λίγο να χτενίσουμε μια κοινή θέση των πολιτικών μας ομάδων όσον αφορά το θέμα αυτό. Συμφωνώ ε, με πολλούς ε, ε, που λένε ότι η γλυφοσάτη δεν είναι ένας αυτός σκοπός, οπωσδήποτε δεν είναι ανώδυνο προϊόν, όπως δεν είναι ανώδυνα και τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε και τον καθαρισμό του σπιτιού. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε πλήρη ανεξαρτησία απέναντι στη βιομηχανία, ένα, και δύο ανεξάρτητες μελέτες έτσι ώστε ε, με, με τα λόγου γνώσεως και έχοντας όλα τα στοιχεία ανεξάρτητα να μπορέσουμε να πάρουμε την τελική απόφαση. Κυρία Γκέρλινγκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα προσπαθήσω να μην μιλήσω πάρα πολύ ώρα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να εξετάσουμε τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Και ναι, βρισκόμαστε και πάλι στην κατάσταση, στην Επιτροπή όπου συζητάμε ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να αποφασιστεί επί επιστημονικών τεκμηρίων και φαίνεται ότι το ξεπετάμε και το τελικά ακούμε συναισθηματισμούς. Ε, θέλουμε λοιπόν να είμαστε και λογικοί και αναλογικοί σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα και τα μέλη της Επιτροπής μιλούν και παίρνουν το λόγο ξανά και ξανά και ε, παρουσιάζουν όχι ε, άκλοντα επιχειρήματα, αλλά προσωπικές απόψεις. Αρνείται η Επιτροπή να αναγνωρίσει τα επιστημονικά απορίσματα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και αυτό με ενοχλεί. Άρα, μιλάμε για τις εφαρμοστικές ε, ιδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν βλέπω όμως σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, γιατί κατά πόσον εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης ή όχι. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι την παραβιάζουμε, γιατί τι λέει η αρχή της πρόληψης. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος, όχι, αλλά ότι εισηγίζουμε τα υπέρ και τα κατά. Αυτό κάνουμε λοιπόν. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο ή λογικό να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τα επιστημονικά τεκμήρια και τις ε, έρευνες. Ήταν σαφές την προηγούμενη εβδομάδα στην παρουσίαση, το κάνανε αυτό και Πώς γίνεται δύο άτομα να ακούν την ίδια παρουσίαση και να καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα αυτό. Θα πρέπει να το φιλτράρουμε ως πολιτικοί. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θεωρώ ότι είναι πραγματικά και παράλογο αλλά και άδικο να πούμε ότι η ΕΚΑ και η ΕΦΣΑ δεν έχουν εξετάσει και δεν έχουν λάβει υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία. Θεωρώ ότι το έχουν κάνει και θεωρώ ότι με σωστού ε, συλλογισμού προτείνουν την ανανέωση για 10 χρόνια τώρα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το σχέδιο. Μιλάμε για το άρθρο 4. Αναφέρεται το άρθρο 4 και ότι δεν συνάδει με, τη βιώσιμη, με την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση. Οι γενικές αρχές για την συνολική διαχείριση των παρασύτων αναφέρονται εδώ. Και φαίνεται ότι όσοι υποστηρίζουν τις απόψεις αυτές δεν έχουν διαβάσει τις γενικές αυτές αρχές για την γενική διαχείριση, τη συνολική διαχείριση των παρασύτων. Αλλιώ δεν θα έλεγαν αυτά που λένε. Έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παράταση για 7 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα έκτοτε και παρόλα αυτά τα μέλη λένε ότι πρέπει να μειωθεί αυτή η περίοδο σε 3 έτη και θα πρέπει να υπάρχει σταδιακή κατάργηση σε 3 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όμω από τότε που πριν από κάποιο καιρό, ε, λίγο καιρό. Ε, ψηφίσαμε το ψήφισμα αυτό. Θεωρώ ότι θα κάνετε περίγελο το Κοινοβούλιο αν υποστηρίζετε τέτοια στοιχεία και μου κάνει εντύπωση αυτό που αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιφρονεί τον ευρωπαϊκό λαό και μιλάτε για ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύριο ανθρώπους. Τι ποσοστό είναι αυτό της συνολικών κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προσυπογράψει δηλαδή μία αίτηση η οποία θα αλλάξει τον τρόπο εργασία μας και ζωή μας. Ε, όχι, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με, αλλά είμαι η πρώτη που μιλάει σε ό,τι αφορά αυτή την πλευρά του ψηφίσματα. Ε, επί μισής ώρας ε, ε, για μισή ώρα ακούμε άτομα τα οποία υποστηρίζουν το ψήφισμα. Είμαι η πρώτη που μιλάει κατά του ψηφίσματο αυτό. Ναι, λέει η πρόεδρο, σα παρακαλώ, προσπαθείτε να περιοριστείτε. Ναι, είμαι σε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά έχω μιλήσει. Όχι, λέει η πρόεδρο, απλά διευκρινίζω. Ναι, προσπαθώ, προσπαθώ. Αλλά έχω και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θέλω να σα παρουσιάσω. Θα ήθελα να υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό την έκκληση για ανεξάρτητε έρευνε εφόσον συνάδουν με τις καλές πρακτικές καλές εργαστηριακές πρακτικές και τις, ε, τα διεθνή πρότυπα τα σχετικά. Επίσης, σύμφωνο ότι θα πρέπει να υπάρξει επαρκή ε, δικασία για δοκιμές και για εξέβρεση ασφαλιστικών δικλείδων. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί αποτελεί συνήθεια πρακτική. Και θα πρέπει να το προωθήσουμε. Αλλά η ιδέα που προβάλλεται από τους υποστηρικτές του αιτήματο ότι υπάρχει μεγάλη και μαζική ανησυχία για την κλεφοσάτη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά τέτοια ανησυχία, αλλά δεν πιστεύω αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 10 για την πρόταση τη ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαχθούν σταδιακά μέτρα κατάργηση της γλυφωσάτης και για την δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών για χαμηλότερε ε, κινδύνου εναλλακτικέ αποτελεί ε, κάτι που περιλαμβάνεται στην ΚΑΠ. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που απονοείται εδώ πέρα στο ψήφισμα, ότι ε, εμπλέκεται η κοινή αγροτική πολιτική. Άρα, καλό είναι ως πολιτική δήλωση, αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε πολύ χρόνο στην Επιτροπή. Αλλά συγγνώμη, εσείς το βάλετε το ψήφισμα. Έχετε τουλάχιστον καθήκον να ακούσετε αυτούς που είναι αντίθετοι. Αλλά συνεψίζοντας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορώ να υποστηρίξω, αλλά πραγματικά είμαι πραγματικά υπέρ συνολικά της ανανέωσης της έγκρισης της γλυφοσάτης. Ελπίζω τέτοια απόφαση να λάβουν τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους ομιλητές. Αρκετά μακροσκελής κατάλογος. Ο κύριος Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να φτιάξω μια γέφυρα και το είπε και η κυρία Αντελάη πριν από λίγο. Εμείς ως ΕΛΚ σήμερα δεν θα υποστηρίξουμε στη φάση αυτή το ψήφισμα. Γιατί θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δρά με συνοχή, να ενεργεί με συνοχή. Πέρσι ψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα. Και σε αυτό αναφέρθηκε μια ετή περίοδος. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο 1,5 χρόνο, είναι η θέση της ΕΚΑ, την οποία τότε δεν είχαμε στην διάθεσή μας. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της γλυφωσάτης, θεωρείται ότι είναι περιορισμένος. Παρά όλα αυτά, η πολιτική πραγματικότητα, ακόμα και αν το 1,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν αποτελούν σημαντικό ποσοστό της ε, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μία λύση σε βάθος χρόνου, αλλά Τώρα, σταδιακή κατάργηση μέσα σε τρία χρόνια, το να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι αυτό αντίκειται και είναι αντιφατικό με αυτά που έχει ήδη αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην τοποθέτησή μας. Γιατί σε αντίθεση με το Υπουργικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχουμε μια θέση θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ενδεχομένως στα πέντε χρόνια, το τρία ούτε επτά και είμαστε υπέρ αυστηρών ε, προτύπων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, για παράδειγμα, χορήγηση γλυφοσάτη πριν από την ε, σοδιά για να βελτιωθεί ο όγκος της οδείας. Αυτό είναι απαράδεκτο και αυτό μπορούμε κατευθείαν να το απαγορεύσουμε και θα ήθελα λοιπόν επί της βάσης αυτής την οποία δημιουργήσαμε την πριν από 1,5 χρόνο να βρούμε μια ευρεία συνένεση την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια και πραγματικά θα ήθελα να μας εισακούσει στο σημείο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να καταβάλει πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι να επιμένει στα 10 χρόνια τα οποία προτείνει με πολύ περιορισμένου περιορισμού. Νομίζω ότι έτσι δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Ευχαριστώ κύριε Μόζα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνική. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να αρχίσει επιπλέον να, επιτέλους ε, να ακούει ε, τα όσα εμείς έχουμε υποβάλει. Έφτασε η στιγμή που η Κομισιόν, λέω, θα πρέπει να ε, ακούει αυτά που λέμε εμείς ε, και ε, στο παρελθόν. Έχουμε ήδη εκφράσει άποψη επί του θέματος αυτού και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ σωστοί όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα phasing out, μία περίοδος. Το είχαμε πει και τότε, αλλά δεν μας άκουσε η Κομισιόν. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός της χρήσης της γλυφωσάτης ως ακόμα και πριν από την συγκομιδή. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε πλειοψηφία για το ψήφισμα και ευελπιστούμε ότι η Κομισιόν όσον αφορά την γλυφωσάτη θα αλλάξει τελείω πορεία. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το εξή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Γκέρλιν. Θα πρέπει να δρούμε βάσει επιστημονικών τεκμηρίων. Φυσικά όλε οι μελέτε ε, οι οποίε χρηματοδοτούνται από τη Μοντσάτο είναι ύποπτε ε, αλλά δεν έχουμε μόνο και την ΕΦΣΑ, αλλά έχουμε και την, Ευρωπα... την Γερμανική Υπηρεσία για την Αξιολόγηση Κινδύνου, που είναι ανεξάρτητο όργανο. Νομίζω ότι αυτούς μπορούμε να τους ακούσουμε. Σε ό,τι αφορά το, το κατά πόσο είναι καρκινογόνος η ουσία, εδώ αναφέρεται ότι μέσα στη χρήση δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι και ο εμπλουτισμό σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν μακροπρόθεσμα καλό θα ήταν να βρούμε ανακτική λύση για την κλειφοσάτη. Αλλά ζήτησα το λόγο για να τονίσω κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Δεν μιλάμε μόνο για τη γεωργία. Γιατί εκεί μπορούμε να πούμε ότι εκεί υπάρχει και κάποια διαφωνία για το τι είναι καλύτερο. Αυτό α μην το συζητήσουμε καν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά βασικά τίθεται και το θέμα των συντριδρόμων. Αυτό δεν το ανέφερε κανένας, γιατί και εκεί χρησιμοποιείται γλυφοσάτη. Ξέρετε ότι αν σταματήσει η χρήση της γλυφοσάτης, ε, το SNCF, οι Γαλλική συνδεδάδρομοι βρήκαν άλλη ουσία, πολύ πιο τοξική όμως, αν ε, χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος Το ανώβερο από όπου και προέρχομαι σε ό,τι αφορά τη χρήση στην ε, τοπικές γραμμές την απαγορεύσαμε και τελικά διακυβεύθηκε η ασφάλεια η συνδρομική. Θέλουμε φυσικά να συνεχίσει να υπάρχει ο συντρόδρομος, γιατί είναι και φιλικός προς το περιβάλλον. Συζήτησα λοιπόν με τους ηθήνοντες τους πολιτικούς και τους είπα γιατί δεν βγαίνουν να το πούν αυτό. Μας είπαν ότι κοιτάξτε, ε, ισχύει αυτό, αλλά ε, πολλοί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το γλυφοσάτι στον τομέα των μεταφορών. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δική μου περιφέρεια. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε λοιπόν ότι δεν μιλάμε μόνο για τη γεωργία, αλλά μιλάμε και για τους σιδηροδρόμους. Και οι σιδηροδρόμοι χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να βρουν εναλλακτική ουσία και να τα χρησιμοποιήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Η κυρία Γκροστέτ, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική γιατί με κάλυψαν σε πολλά συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να αποκρισταλώσουμε τη γνώμη μας γιατί ακούμε πολλές και διάφορες απόψεις και μετά τη δημόσια ακρόαση αντί να διαλευκανθούν κάποια πράγματα ε, βρεθήκαμε σε μεγαλύτερη ακόμη σύγχυση. Ε, έγιναν κάποιες ε, ε, επισημάσεις για δυνητικούς κινδύνους αλλά ή ούτε οι οργανισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την ε, ε, Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ελβετία, την ΕΦΣΑ, την ΕΧΑ. Ε, δεν υπάρχει παρόλα αυτά, παρά τις πολυάριθμες μελέτες, μια κοινή γραμμή και κοινά συμπεράσματα. Γι' αυτό ζητούμε έντονα ανεξάρτητες μελέτες. Υπάρχουν όμως ανεξάρτητες μελέτες, είναι δυνατόν να έχουμε ανεξάρτητες μελέτες, γιατί και από όποια πλευρά και να τα δούμε τα πράγματα, υπάρχουν πάντα αμφιβολίες. Ε, όπως είπε ο Δ. Λίζα, ίσως θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές ε, και τους όρους για τους οποίους έχουμε συμφωνήσει την άνοιξη του 2016. Ευχαριστώ κυρία Χάζακαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα εκ νέου έχει την ευκαιρία να εισακούσει την έκκληση 1,3 εκατομμυρίων πολιτών για την απαγόρευση της εγλυφωσάτης. Το αντίθετο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με κάθε τίμημα θέλει να παραμείνει στην αγορά. Η δεν ακούει τους πολίτες και δεν ακούει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει βασικά τον παραγωγό δηλητηρίου, τη Μοντσάντο. Κάποιοι λένε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι μπορούμε να παραμείνουμε στην παλιά μα απόφαση. Αυτό δεν αληθεύει όμω, Πρόεδρε, δεν ισχύει. Έχουμε κάνει και μια κρέωση για τα έγγραφα Μοντσάντο και πραγματικά άλλαξε κάτι την τελευταία περίοδο. Πλέον ξέρουμε ότι η Μοντσάντο δεν ε, φύγεται κανένας μέτρου για να προωθήσει το προϊόν αυτό στην αγορά και μάλιστα και από έρευνες δημοσιεύει. Είναι λοιπόν ακατανόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ακούει τη Μοντσάντο. Είναι επικίνδυνο λοιπόν αυτό για τους ανθρώπους, για τα ζώα. Ε, είναι πραγματικά μοιραίο για το περιβάλλον και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φύγει από την αγορά. Εγώ αυτό που προτιμώ είναι τα τρία χρόνια προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν όλοι και οι αγρότες και οι πολίτες και οι πολιτικοί. Ευχαριστώ. Κύριε Σαμαρτζή. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι. Απλώς άκουσα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει. Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει τίποτα. Εμείς απλώς γνωμοδοτούμε για ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και που απασχολεί 1,3 εκατομμύρια συμπολίτε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό όντω δημιουργεί πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Γιατί για ένα τόσο σημαντικό θέμα υγείας και για πολύ σημαντικά θέματα συνενοχής μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των βιομηχανικών λόμπι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία καταστρατηγείται και φύγεται. Νομίζω ότι είναι και η ώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει να δηλιάζει μπροστά στα βιομηχανικά λόμπι, γιατί ε, θα μας ε, φέρουν ενώπιον των ευθυνών μας κάποια στιγμή για κάτι που μπορεί να γίνεται πιο σοβαρά σκάνδαλα υγειονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ε, την ε, Διευθύντρια, ε, τον Διευθυντή, τη Διευθύντρια Γιουλή Κάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνει να σας παρουσιάσουμε τη θέση μας επί του κειμένου του σχεδίου εστάσεων και να απαντήσουμε στα πολύ κατηγορηματικά σχόλια που έγιναν. Καταρχήν, τον Ιούλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στα κράτη-μέλη την πρότασή της για μια εκτελεστική πράξη που εφαρμόζει ουστικά υπάρχοντα κανονισμό έναν κανονισμό που έχει εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτελεστική πράξη λοιπόν για την ανανέωση της έγκριση για την γλυφοσάτη για μία δεκαετία. Και συζητήσαμε την πρότασή μας με τα κράτη-μέλη την τελευταία φορά στις 5 Οκτωβρίου. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόταση αυτή δεν εστάλει ούτε στο Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο ε, σε διαφορετικές ε, στιγμές ε, φορτώθηκε στο Μητρό Επιτροπολογίας στην κατάλληλη στιγμή και τέθηκε αμέσως στη διάθεση των δύο θεσμικών οργάνων. Πρόκειται όντω για ένα ντοσχέ που προκαλεί ζωηρό ενδιαφέρον και από την κοινή γνώμη και μάλιστα στο, στην ιστοσελίδα είχαμε ε, από την αρχή παρουσίαση όλων των ε, γράφων και των αποτελεσμάτων τη συζήτηση. Η πρόταση για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφωσάτη εδράζεται σε ξεκάθαρα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τα συμπεράσματα αυτά συγκεντρώθηκαν μετά από μια πολύ διεξοδική επιστημονική μελέτη της ουσίας αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ αυστηρά κριτήρια για την έγκριση που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη χρήση των ε, ζυζανιοκτώνων και των ενδομοκτώνων. Και μάλιστα ελέγξαν υπόψη και αξιολογήσει Ευρω... του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Τροφίμων για την ταξινόμηση τη γλυφωσάτη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε ω προ πιθανή ε, καρκινογόνο δράση τη ουσία. Και όντω αυτό το αυτό το θέμα ήταν διαφορετικό το 2016 όταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα για την παράταση της έγκρισης της ε, γλυφοσάτης για μία πτέτεια. Έκτοτε έχουμε την επιπλέον επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων που είναι κατά της ε, ταξινόμης της γλυφοσάτης ως καρκινογόνου ουσίας. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την ανανέωση αυτή ε, ευθυγραμμίζεται πλήρω με τι διαδικασίε και του όρου για την ε, παροχή των ε, δεδομένων, την παραγωγή των δεδομένων και από τον ετώντα την διαφάνεια και την επιστημονική αξιολόγηση όπως προβλέπεται από την τρέχουσα ενωσιακή νομοθεσία που εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ακούσαμε κάποιους ισχυρισμούς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοφεύει υποτίθεται θα ήθελα να σα επισημάνω ότι η πρόταση για την ανανέωση τη γλυφωσάτη λαμβάνει υπόψη και άλλου θεμητού παράγοντε. Για παράδειγμα το ψήφισμά σα του Απριλίου του 2016. Εκεί ζητάτε ε, μια επταετή ανανέωση τη άδεια και την ε, πρωτοβουλία των πολιτών που επισήμω ε, υπευλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Οκτωβρίου του Τρέχοντο έτου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια περίοδο ανανόηση 10 ετών και όχι την ε, μέγιστη περίοδο ανανέωση που προβλέπετε των 15 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες ε, και αυτούς τους θεμητούς παράγοντες. Τώρα, απαντώντας σε κάποιες ε, παραγράφους του ψηφίσματος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η διεξοδική και περιστατωμένη μελέτη όλων των στοιχείων δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος η γλυφοσάτη. Επίσης, η ομάδα εκτιμηση κινδύνου του ΕΧΑ και της ΕΦΣΑ με υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί καρκινογόνος ή γλυφοσάτη. Επίσης, η συζήτηση για επιστημονικά στοιχεία, απορίσματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις ε, σε μια σύντομη συζήτηση όπως αυτή που έγινε εδώ σήμερα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια διεξοδική και περιστατωμένη επιστημονική διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, η γνωμοδότηση των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών, του ΕΧΑ και του ΕΦΣΑ, που άλλωστε υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και που θεωρούν ότι η γλυφοσάτη δεν θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, γίνεται δεκτή και από άλλους φορείς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλούμε για ε, έγκυρες και κορυφαίους αρχές και φορείς της ε, Νέας Ζηλανδίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά και ούτω καθεξής. Και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας άλλωστε, και οι φορείς του που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Είχαμε την κοινή συνάντηση για τα κατάλοιπα των εντομοκτώνων που κατέληξαν επίσης τα ίδια συμπεράσματα. Οπότε μόνο ένας φορέας του ΠΟΗ έχει διαφορετική γνώμη για το θέμα αυτό και είναι πραγματικά μεμονωμένη αυτή η άποψη. Οπότε, εν κατακλείδη, το θέμα του κατά πόσο η γλυφοσάτη προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο, το θέμα αυτό έχει απαντηθεί με ικανοποιητικό κατά τη γνώμη μας τρόπο. Ε, βέβαια, μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλοι φορεί προσπαθούν να απαξιώσουν αυτή την επιστημονική αξιολόγηση που έγινε για τη γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από του ευρωπαϊκού οργανισμού ΕΧΑ και ΕΦΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη ισχυρισμού, ακόμη και μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των ισχυρισμών που ακούσαμε και στην πρωινή συζήτηση και γι' αυτό ε, συνεχίζουμε να ζητούμε από τους διοργανισμούς ε, να μελετήσουν το θέμα Προσπαθώντα να απαντήσει στους ισχυρισμού που έγιναν για την γλυφοσάτη. Σας διαβεβαιώ ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνε μας. Και όπως θα διαπιστώσατε από τις δηλώσεις των δύο οργανισμών και από το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκτιμήσεω Κινδύνου, έγινε μια διαφανής διαδικασία και η ευρωπαϊκή διαδικασία ε, για, την, ε, για τα εντομοκτώνα εφαρμόστηκε και στη γλυφοσάτη με διαφάνεια. Νομίζω ότι οι αμφιβολίες κανονικά θα έπρεπε να διασκεδαστούν μετά από τη διαφανή αυτή διαδικασία και μετά από τα πορίσματα αυτών των δύο ανεξάρτητων ενωσιακών οργανισμών που απεφάνθησαν κατά του καρκινοβόρου χαρακτήρα της γλυφοσάτης. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση που υπευλήθη στα κράτη-μέλη εδράζεται σε έγκυρα επιστημονικά πορίσματα μετά από διεξοδικό ε, και εμπεριστατωμένο έλεγχο και από τα κράτη-μέλη και από τους εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, υπάρχει λόγος για να τεθούν ένα φιβόλο αυτά τα συμπεράσματα για τη γλυφοσάτη. Και μια και α, ε, τηρήσαμε τις α, κανονιστικές διαδικασίες και μάλιστα σχολαστικά, ε, θεωρώ ότι δεν υπερβαίνουμε τις εκτελεστικές μας ε, αρμοδιότητες κατά την υποβολή της σχετικής πρότασης. Επίσης κάποια άλλα θέματα που επισημάνατε περί διαφάνειας ε, και εδώ θεωρούμε ότι το ισχύον σύστημα όπως έχει αποφασιστεί από τους δύο συνομοθέτες ήδη εφαρμόζει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας με τη δημοσίευση πολλών στοιχείων και πληροφοριών και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Ως προς το θέμα της διαφάνειας λοιπόν, ε, θεωρώ ότι υπάρχουν εξελίξεις, το είδαμε ε, και για τα φάρμακα στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα της διαφάνειας με αλλεπάλληλες αξιολογήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη γενική νομοθεσία των τροφίμων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του REFIT για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα των εντομοκτώνων. Και ζυζανιοκτώνων. Και πλησιάζω προς το τέλος της παρέμβασής μου. Ε, τέθη ένα ερώτημα ε, για το κατά πόσο προτείνουμε την δεκαετή ανανέωση υπό την απειλή για προσφυγή στο δικαστήριο των εταιριών. Όχι, σας διαβεβαιώ, δεν γίνεται υπό την επίρρεια του φόβου αυτή η πρόταση αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα, τις ε, ανησυχίες που επισημάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και προτείναμε δεκαετή και όχι 15 ετή ανανέωση. Επίσης δεν θα λάβω θέση απέναντι στα πολύ κατηγορηματικά σχόλια που έγιναν κατά τη γνώμη μου και πολύ δρυμία κριτική βάρος των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επροκειμένου και κάποιων ευρωπαϊκών οργανισμών, θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι φορείς ακολουθούν πιστά την ενωσιακή νομοθεσία, ε, της και της ε, ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το ψήφισμά σας. Δεν υπάρχουν επιστημονικά πορίσματα για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ το σχέδιο ψηφίσματός σας ε, σε πολλά επιμεροσημεία σημεία μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη στο ενωσιακό σύστημα και στο έργο των ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν επιτελέσει επάξια το έργο τους σε πολλούς άλλους τομείς όπως τα νεόνικοτινοειδή για παράδειγμα. Εκεί οι αρχές μας εξυπηρέτησαν και μας ε, επέτρεψαν να επιτελέσουμε την αποστολή μας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν τρία ψηφίσματα σχετικά με γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα. Ε, δεν έχουμε χρόνο. Διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Ε, έχουν προβλεφθεί ψηφοφορίες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουμε όλοι δεσμεύσεις. Πρέπει οπωσδήποτε οι ψηφοφορίες να λάβουν χώρα την προβλεπόμενη ώρα. Ε, πρόεδρος, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ψηφιστούν αυτές οι ενστάσεις. Εάν όλοι συμφωνήσουν ε, να γίνει ψηφοφορία επί των ενστάσεων αυτών χωρίς συζήτηση, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι το θέμα έχει θυγεί πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει, γνωρίζουμε τα ε, επιχειρήματα. Ποιος θα ήθελε λοιπόν να ψηφίσουμε για τις ενστάσεις επί των γενετικών τροποποιημένων χωρίς συζήτηση. Υπέρ, κατά, αποχές, Εντάξει λοιπόν, άρα συμφωνούμε, άρα μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες και ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκροστέτε για την ε, πρόταση που κάνατε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που την υποστήριξαν. Okay, uh, Ωραία, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε την ε, ε, κάρτα σας Είσαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για την ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία λοιπόν σχετικά με την έσταση για την Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα Κύριε Παρδιό θέλετε κάτι? Όχι. Ένσταση λοιπόν σχετικά με τι προϊόντα τα οποία περιέχουν, περιλαμβάνουν ή παράγονται ε, με ε, ε, σόγια γενετικώς τροποποιημένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. We vote Let's try to keep the voice down. Μη φωνασκείτε παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Ψηφίζουμε ε, για την ε, ένσταση σχετικά ε, με την χρήση γενετικώς τρεποποιημένη ε, ελαιοκράμβη μόνο 88302 άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Έχουμε άλλη μία ένσταση σχετικά με την διοδότηση ε, προϊόντων που περιέχουν ή περιλαμβάνουν τροποποιημένο καλαμπόκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ψήφιση έκθεσης ε, που αφορά την προστασία των εργαζομένων σχετικά με την έκθεσή τους σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρι... Ε, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία όσον αφορά την τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη η έκθεση. Η κυρία Μελίνα έχει ζητήσει το λόγο ναι, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι υπερψήφισαν το θέμα αυτό. Θα ήθελα πάντως να παρατηρήσω ότι για δεύτερη φορά η Επιτροπή μας δεν θα δώσει γνωμοδότηση στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι ε, όταν έχουμε καρκινογόνες ε, ουσίες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα ε, καρκινογόνες θα έπρεπε τουλάχιστον να δώσουμε την ίδια προσοχή με αυτή που δίνουμε στην γλυφοσάτη η οποία δεν είναι αποδεδειγμένα πλήρως καρκινογόνος. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία ε, σχετικά ε, με ε, κείμενο το οποίο αφορά τις, τον τομέα της, του μελιού. Ευχαριστώ ε, πολύ, κυρία Ντοναρό. Θα ήθελα να ε, ζητήσω χωριστή ψηφοφορία ε, για τις 3092 όσον αφορά την έκθεσή μου για τον... τον τομέα της μελισσοκομείας. So για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε τέτοια αίτηση θα πρέπει ε, να σας υποστηρίξουν οι συνάδελφοί σας. Ε, ποιος υποστηρίζει, μάλλον όχι, ηλεκτρονικά να δούμε εάν συμφωνείτε με την πρόταση της κυρίας Ντορνανό. Πέρας. Απερίφθη. Α, όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος διορθώνει, διότι έχετε 18 ε, ψήφους υπέρ ε, όσους χρειάζεστε λοιπόν. Πολύ ωραία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά Η άλλη δεν ψήφισε. να ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, άρα ηλεκτρονικά να το δούμε. Πέρας, εγκρίνεται. Ε, πραγματικά σας βεβαιώ ότι δεν ήταν καθόλου σαφές ε, πριν το αποτέλεσμα. Τροπολογία 10, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 24, τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές. Ξανά. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Καταπίπτουν κάποιες τροπολογίες λοιπόν. Και περνάμε στην τροπολογία 28, ε, έτοιμα ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ξανά όμως να ψηφίσουμε. Ε, τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί ε, της τροπολογίας 46 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ όχι μάλλον θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 47 ωραία ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 47 Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 53 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 54 ε, με ε, ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απερίφθη. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήθελε, όχι, καλύτερα να κάνουμε μια επαλήθευση Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την 69. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 73. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει αυτή. 77. Τροπολογία, όχι, τροπολογία 75 διορθώνει η Πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές. Αμφίβολο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ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 91. 91. 91 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 ε, με ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η κυρία Ντορνανό. Πέρασε. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Αλλά δεν ψήφισε το ΑΕΛΚ, οπότε ξανά, τροπολογία 99, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πάλι δεν έχω εικόνα, λέει η Πρόεδρος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας, τροπολογία 99, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 100, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 105 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της τροπολογίας 105 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Και πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Αυτό είναι πολύ καλό. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Okay. Θα σε προσκαλέσω, αν ε, σκοπεύετε να συμμετάσχετε στην επόμενη συζήτηση, παρακαλώ να καθίσετε. Για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εξελίξεις του ΙΚΑΟ σε ό,τι αφορά το Κόρσια. Τη αντιστάθμιση να ανθέκα και των μείωσης ε, του άνθρακα. We, uh, have... Uh, Και έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μας Έχουμε προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσει το θέμα αυτό μαζί μας. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Πέτρε Βης, σύμβουλο στην Γενική Διεύθυνση μεταφορών και κινητικότητας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω τα μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής σας σε ό,τι αφορά τις ε, εξελίξεις ε, στον ΙΚΑΟ, σε ό,τι αφορά το σύστημα της στάθμισης εκπομπών άνθρακα και προγραμμάτων μείωσης στη διεθνή πολιτική αεροπορία. Ε, κόρσια, εν συντομία, και με την άδειά σας κυρία Πρόεδρε, να σας πω ότι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε σύνοδο του ΙΚΑΟ στο Μεξικό Σίτι για τη βιώσιμη αεροπορία. Στο τέλος όμως της παρουσίασής μου. Το Κόρσια θα εφαρμοστεί μέσω των προτύπων και συστημένων άμα πρακτικών της ΕΚΑΟ το ΣΑΡΠ όπως ονομάζεται. Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και θα τεθεί σε εφαρμογή α, το ΣΑΡΠ και το υποστηρικτικό σύστημα από τις αρχές του 2009. Τα κράτη μπορούν να συμμετέχουν, να συμμετέχουν εθελοντικά στο Κορσία μέχρι τον Ιούνιο του 2020 και κάθε έτος ε, πέρα από το 2020. Το 2027 ξεκινάει η υποχρεωτική περίοδος εφαρμογής από το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, 72 κράτη που εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν 87,7% της ε, διεθνούς ε, δραστηριότητας αεροπορίας ε, είχαν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο Κόρσια από την αρχή του προγράμματος, από το 2021. Και αυτό θα ήταν, είναι η καλύτερη κάλυψη αν είχαμε συμφωνήσει για μια σταδιακή υποχρεωτική η φάση εφαρμογή, όπω είχε στην αρχή προταθεί. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν, για την παράταση τη ε, διαδικασία περίοδου αναστολή ε, stopping the clock, προκειμένου να παραταθεί η εξαίρεση των ε, κρατών τρίτων, των πτήσεων τρίτων χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ETS για περαιτέρω περίοδο, θα ήταν ευπρόσδεκτη, γιατί έτσι θα συνεχίσουν να διευκολύνονται οι συζητήσει για το κόρσια στο ΕΚΑΟ. Η Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό ήθελε ένα μηχανισμό παγκόσμιο βάσει της αγοράς και η Ευρώπη έχει καταβάλει γιατρές προσπάθειες για να ανατηρηθεί η περιβαλλοντική ακαιρεότητα του κόρσια. Το κόρσια είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για να υπάρξει ένας μηχανισμός παγκόσμιος βάσει της αγοράς και να συμπληρωθούν τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται από την ε, διεθνή ε, τομέα πολιτικής αεροπορίας και ως ένας τομέας ο οποίος εξαιρείται, από τις εθνικώς καθορισμένες συνεισφορές της Συμφωνίας του Παρισιού ε, είναι μεγάλη σημασία η διεθνή πολιτική αεροπορία να συνεισφέρει στις προσπάθειες να μειωθεί η θερμοκρασία κατά 1,5 έως 2 βαθμούς και ο διεθνής κλάδος ξέρει τι περιμένουμε από αυτόν. Στην συνάντηση 11-15 Σεπτεμβρίου του 2017 η Διευθυντική Ομάδα της Επιτροπής Προστασίας ε, ε, και Περιβαλλοντικής Προστασίας του ΙΚΑΟ, η ΚΑΠ, συμφώνησε επί ενός πακέτου, ενός σχεδίου πακέτου για το κορσέ το οποίο θα συσταθεί για έγκριση από το Συμβούλιο του ΙΚΑΟ. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει λοιπόν ένα σχέδιο ΣΑΡΣ υποστηρικτικές πληροφορίες και τεκμηρίωση και ένα περιβαλλοντικό τεχνικό εγχειρίδιο. Το ΚΕΙΠ αποτελεί λοιπόν ένα συμβουλευτικό σώμα προς το Συμβούλιο ΙΚΑΟ και ε, εγώ είμαι εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΚΕΙΠ και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παρατηρητή και όχι πλήρες μέλος, δίνουμε παρόλα αυτά τη συνεισφορά μας στις ε, διαβουλεύσεις του ΚΕΙΠ τα ευρωπαϊκά κράτη θεωρούν ότι το πακέτο Κόρσια αντιπροσωπεύει ένα μ, ικανοποιητικό πακέτο. Η ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τους Ευρωπαίους συμπραγματευτές στην ακαιριότητα των κριτήριων για τις μονάδες εκπομπών και την βιωσιμότητα και τα κριτήρια βιωσιμότητας για εναλλακτικά καύσιμα, βιώσιμα καύσιμα και εστιαζόμαστε στους τρεις πυλώνες της ε, βιωσιμότητας, ο περιφερειακός, κοινωνικός και οικονομικός πυλώνας. Πριν τις περαιτέρω του Συμβουλίου του ΙΚΕΟ θα δοθούν ε, και συνεισφορές από δύο άλλα σώματα, το συμβουλευτικό, η συμβουλευτική ομάδα για το κόσια και την ε, ομάδα πλοήγησης του ΙΚΑΟ. Το Συμβούλιο του ΙΚΑΟ θα συνδεθεί στις 30 Οκτωβρίου του 2017 μέχρι 17 Νοεμβρίου του 2017 και αναμένεται ότι θα αποφασίσει επί του πακέτου Κόρσια, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στα κράτη για σχολιασμό. Η τελική δε έγκριση αναμένεται για τον Ιούνιο του 2018, προκειμένου τα ΣΑΠΣ και οι υποστηρικτικές πληροφορίες να ξεκινήσουν να ισχύουν από την αρχή του 2019. Και κατά τη διάρκεια του 2018 οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει να υποβάλουν ε, λεπτομερή σχέδια για το πώ θα παρακολουθούν και θα χορηγούν προ έγκριση την κατανάλωση καυσίμων του για το 2019 και 2020. Όλα τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στην διεθνή αεροπλοεία θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αεροπορικέ εταιρείε θα καταγράφουν τι εκπομπέ από την διεθνή αεροπλοεία. Αυτό είναι πάρα πολύ στενό χρονικό διάστημα και χρονικό περιθώριο και θα προαπαιτήσει πολύ σημαντικές προσπάθειες από τις εταιρείες οι οποίες ενδεχομένω να μην έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα. Αυτά τα αναφέρω για να τονίσω την τεράστια παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται και από τα κράτη τα οποία ενδεχομένω δεν έχουν οπτήν για την εθελοντική φάση του Κόρσια. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη του Κόρσια. Την επόμενη εβδομάδα οι τεχνικοί εμπειρογνώμονε θα συναντηθούν στη Βραζιλία για να αναπτύξουν περαιτέρω τεχνικέ λεπτομέρειε που δεν χρειάζονται ενδεχομένω στο πακέτο του Κόρσια το καθεαυτό, αλλά θα χρειαστούν στη φάση πρακτική υλοποίηση εφαρμογή του Κόρσια. Και η εργασία αυτή θα εστιαστεί σε λειτουργίε καταχώρηση, σε ένα απλοποιημένο εργαλείο αναφορά και περαιτέρω δουλειά για τα βιώσιμα καύσιμα εναλλακτικά καύσιμα. Θα εστιατούμε δηλαδή κυρίω στην υλοποίηση και την εφαρμογή και όχι τόσο στο το μέσο. Ο βασικό σχεδιασμό έχει ολοκληρωθεί, αλλά χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των λεπτομεριών. Επίση, να αναφέρουμε ότι ενδεχομένω το Κόρσια να εξελιχθεί στην, με την πάροδο του χρόνου μέσω των αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων από τους ε, εμπειρογνώμονες. Η πρώτη αναθεώρηση θα λάβει χώρα το 2022. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, στο Μεξικό City την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα η δεύτερη διάσκεψη του ΙΚΑΟ για τα εναλλακτικά καύσιμα αεροπορίας και εγκρίθηκε μία δήλωση η οποία αναφέρει τα εξή. Η διάσκεψη αναγνωρίζει ότι η βιωσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων αεροπλοεία είναι κρίσιμη σημασία για τι προσπάθειε τη διεθνού αεροπλοεία να μειώσει τι εκπομπέ διεξοδίτου του Αυτό εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα καύσιμα αεροπλοεία, όπω εξετάζονται στην παρούσα φάση από το ΕΚΑΟ. Δεν εγκρίθηκαν ποσοτικοί στόχοι στη διάσκεψη σε αφορά την χρήση των βιώσιμων καυσίμων, αλλά αναγνωρίζεται με σαφήνεια ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερε προσπάθειε και ότι τα βιώσιμα καύσιμα τη αεροπορία, στην αεροπορία μπορούν ε, να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών της διεθνούς αεροπορίας και το επίτευγμα των τελευταίων μηνών είναι ότι τα βιώσιμα αυτά καύσιμα έχουν μπει στο επίκεντρο των προσπαθειών των μελλοντικών σε ό,τι αφορά την πολιτική αεροπορία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε και είμαστε και εγώ και η ομάδα μου στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τα ενδεχομένως έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βίσ. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Πίτερ Βίς για την ενημέρωση που μας έκανε. Έχω μερικές απορίες. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η κόρση αντιστάθμιση κομπών και προγράμματο μείωση στη διεθνή πολιτική αεροπορία. Γι' αυτό όλοι συμφωνούμε. Έχω μερικές ερωτήσεις. Μερικές μπορεί να είναι ρητορικέ, αλλά ε, επειδή ε, είμαστε απασχολημένοι στο τριμερή διάλογο, δεν ε, ε, μείναμε ενήμεροι με τις τελευταίες εξελίξεις όπως προκύπτουν από την ιστοσελίδα σας. Ποιες είναι οι συστάσεις της ΚΑΠ, της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο της ε, ΚΑΟ και είναι προσιτές στο κοινό. Γιατί αν δεν είναι δημόσια σε αυτές οι συστάσεις της ΚΑΕΠ υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας. Και... Είπατε ότι πριν τη συζήτηση δεν θα υπήρχαν, αλλά τώρα είναι ε, προσβάσιμες οι πληροφορίες αυτές, οι συστάσεις της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, της ΚΑΕΠ. Είπατε ότι ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή αυτή την ΚΑΕΠ ε, φροντίζεται να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του Κόρσια της αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα. Μπορείτε να μας πείτε δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσετε. πώς έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά την διαφύλαξη της ε, περιβαλλοντικής ακαιρεότητας ε, στις συστάσεις της ΚΑΕΠ. Πώς έχουμε προχωρήσει, έχουμε εξασφαλίσει αυτή την ισορροπία για να προφυλάξουμε αυτή την ακαιρεότητα την περιβαλλοντική. Επίσης, ε, το 2019-2020 ξεκινά να λειτουργεί το MRV. Και αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και ιδιαίτερα ε, στις ε, τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν δεν μπήκαν και θελώς στην πιλωτική φάση. Οι εταιρείε που δεν έχουν μπει σε αυτή την πιλωτική φάση, αλλά είναι μέλη της ΕΚΑΟ θα εφαρμόσουν διαδικασίες MRV στην πιλωτική φάση, άσχετα από το αν ε, έχουν ε, ενταχθεί θελοντικά ή όχι. Ο κύριος Σελίζ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βίς για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Θα ήθελα, επειδή έγινε χθε το βράδυ, να πω συγχαρητήρια στην κυρία Βαλεάν και στην κυρία Γκέρλινγκ ότι πετύχαμε χθε τη συμφωνία να κάνουμε αναστολή της περίοδου αυτή, το stop the clock. Δεν είμαι 100% ικανοποιημένος, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε ένα συμβιβασμό το ανθεντικό αυτό. Και μέχρι το 2023 θα υπάρχει το σύστημα το ευρωπαϊκό, το ETS, ε, αλλά και πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση σε ό,τι αφορά την πλήρη ε, εφαρμογή. Δείχνουμε λοιπόν μία ένδειξη καλή θέληση προ τον ΙΚΑΟ, αλλά θέλουμε να ασκήσουμε και πίεση παράλληλα. Λέγοντα ότι αν η συμφωνία είναι κενή και δεν βοηθήσει καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένω η Ευρώπη να επιβάλλει το ETS, το σύστημα εμπορία ρήπων και σε τρίτε χώρε. Να θίξω λοιπόν ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να μας δώσει και μια σαφή κατεύθυνση για τις διαπραγματεύσεις. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα των αντισταθμίσεων των offsets. Στην Ευρώπη καταργήσαμε τις αντισταθμίσεις με τις αποφάσεις που λάβαμε σχετικά με το σύστημα εμπορίας λοιπόν το ETS, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην βρεθούμε με τα ίδια προβλήματα στον ΙΚΑΟ που είχαμε στην Ευρώπη. Κακής ποιότητος offsets, ε, αντισταθμίσεις και κάτι με προβλημάτισε, να σας πω την αλήθεια. Σοβαροί εκπρόσωποι αεροπορικών εταιριών ε, στην Ευρώπη μας δήλωσαν ότι φυσικά δεν πρόκειται να φυτέψουμε δέντρα, γιατί αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Αλλά στην διάσκεψη του κλίματος ακούσαμε από τη Γενική Διευθύντρια του ΙΚΑΟ, είδαμε ένα βίντεο ότι να φυτεύουμε φυτά, φυτεύουμε δέντρα και αυτό αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα αντισταθμίσεων θα ήθελα να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ρεαλιστικό να καταργηθούν αυτά τα πολύ αμφιλεγόμενα μέτρα αντισταθμίσεων. Τέλος, κάτι θετικό, γιατί χρειάζεται και λίγο ελπίδα σε όλο το δίλημα αυτό, γιατί προφανώς όλοι θέλουμε να χρησιμοποιούμε αεροπορικές πτήσεις, αλλά αν συνεχιστούν τα πράγματα όσα έχουν σήμερα, οι πτήσεις θα αποτελέσουν το βασικό πρόβλημα για το κλίμα. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που είναι πολύ πιστικό στην διάσκεψη για το κλίμα είναι ότι οι εκπρόσωποι του ΙΚΑ έχουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το πώς θα μπορεί κανείς να πετάει με ουδέτερο τρόπο. Φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, τεχνολογίες χερσαίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και βιώσιμα βιοκαύσιμα. Θα ψηφίσουμε την άλλη Δευτέρα την έκθεση του Μπασάικα του το θέμα αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές πτήσεις και τις μεταφορές αυτές. Ε, ένα τμήμα να χρησιμοποιείται για με βιώσιμα τέτοια καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν τα βιώσιμα αυτά καύσιμα να τα χρησιμοποιούμε όλα 100% στις ε, οδικές μεταφορές και να μην μένει τίποτα για την αεροπορία. Και θεωρώ ότι είναι καλά αυτά τα οποία συμφώνησα με του κοιόδους ο Μπάς Άικαουτ. Αλλά να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτίθεται να ακολουθήσει αυτή την πρόταση γιατί θεωρούμε ότι δεν δίνονται επαρκή κίνητρα στον οικονομικό κλάδο προκειμένου να διαθέσουν και στην αεροπορία σε επαρκέ ποσοστό τέτοια βιώσιμα καύσιμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση, πολύ σημαντική και είμαι απόλυτα πεπισμένη μετά τις τελευταίες εξελίξεις ε, ότι το Κόρσια μπορεί να σταθεί με επιτυχία, να αποτελέσει απόλυτη επιτυχία και μετά το Παρίσι και μετά τις υπόλοιπες διασκέψεις για το κλίμα θα έπρεπε να συμμετάσχει στο βαθμό του δυνατού όλος ο κόσμος, 70% δηλαδή των κρατών, 90% των συνολικών εκπομπών είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαι αισιόδοξη, πάντα ξέρετε, πολλοί ασχολούνται και με εναλλακτικά υλικά, εναλλακτικά καύσιμα για την αεροπορία, αλλά ένα άλλο σημαντικό σκέλος είναι και πιο ελαφριά υλικά για την αεροπορία. Και υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ ε, ιδέες σε ό,τι αφορά τη χρήση πιο ελαφριών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι μιλήσατε για εναλλακτικά καύσιμα. Αναφέρατε συγκεκριμένα ζητήματα. Ε, τι γίνεται για παράδειγμα με τις περιπτώσεις ε, παραμονής στα αεροδρόμια. Τι γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού στα αεροδρόμια, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη χρήση α, άλγης για την ηλεκτροδότηση στα αεροδρόμια και για άλλε περιπτώσει. Κυρία Ντάρλινγκ. Κυρία Ντάρλινγκ, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ε, τον Πίτερ Βις για την ενημέρωση. Μπράβο σας για τη συμφωνία Stop the Clock ε, που συνήθει χθε. Όντως, ε, οι φορείς αυτοί στέλνουν θετικά μηνύματα προς, την, προς τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τη Συμφωνία των Παρισίων, γιατί ε, επιμένουμε ότι η Συμφωνία των Παρισίων απαιτεί δράσεις από όλους τους φορείς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και είναι γνωστό ότι η διεθνής ε, ε, αεροπορία δεν Ξέρετε από τη συμφωνία αυτή. Αυτό το τονίσαμε και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το έχει τονίσει και η ίδια η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα θα πρέπει η ΚΑΟ να αποδείξει ότι είναι ε, προορατικό ε, φορέας, και ε, παράγοντα. μπορεί να προτείνει μέτρα που θα εφαρμοστούν εύκολα από τον κλάδο για να σηματοδοτήσουν μια πραγματική διαφορά και πρόοδο. Και Χαίρομαι για πρωτοβουλίες και μέτρα που θέλει να αναλάβει η ΚΑΟ, αλλά πώς ε, θα μεριμνήσουμε ώστε τα αποτελέσματα της ΙΚΑΟ ε, ε, να εξασφαλίσουν όντως βιώσιμη ανάπτυξη της αεροπορίας, μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και συμβολή, συνεισφορά και της ΕΚΑΟ στις παγκόσμιες προσπάθειες για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Θέλουμε οι προσπάθειες της ΕΚΑΟ να είναι αξιόπιστες, ρεαλιστικές και κυρίως να έχουν ε, απτά αποτελέσματα, να επιφέρουν δηλαδή ουσιαστικές ε, ε, και ορατές αλλαγές. Συμβαίνει αυτό. Επίσης, τι κατεύθυνση ακολουθεί η ΕΚΑΟ σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα. Ε, έχει ένα στόχο 2% βιοκαύσιμα για την αεροπορία μέχρι το 2025 και θα με διέφεραν οι απόψεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της ΕΚΑΟ για τα βιοκαύσιμα. Δεν έχω άλλους ε, ομιλητές στον κατάλογο, δεν ξέρω αν παρέλειψα κάποιον, θέλει να προσθεθεί κάποιος στον κατάλογο, όχι. Οπότε επιστρέφουμε στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πέτερ Βίση, για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα βάλω τα δυνατά μου για να απαντήσω. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκέρλινγκ για το κατά πόσο α, ε, οι συστάσει της ΚΑΕΠ στο Συμβούλιο της ΙΚΑΟ είναι δημοσίως προσβάσιμα. Όχι, δεν είναι δημόσια αυτά τα έγγραφα, ε, αυτές οι συστάσεις της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Και η κυρία Γκέρλινγκ και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, ε, γνωρίζει ενώ και γνωρίζετε ότι η ΚΑΕΠ είναι συμβουλευτική επιτροπή που παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στο Συμβούλιο της ΙΚΑΟ, αλλά οι συζητήσεις της ΚΑΕΠ και τα έγγραφα της ΚΑΕΠ ε, είναι εμπιστευτικά, δεν ε, διατίθενται δημόσια. Βέβαια, στην ΚΑΕΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι και των χωρών, αλλά και των ενδιαφερομένων ε, της βιομηχανίας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οπότε είναι σύνθετη η σύνθεση της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Τώρα, ε, πότε είναι δημόσιες αυτές οι στάσεις. Όταν ε, εγκριθούν και επίσημα τα πρότυπα και οι συνιστόμενες πρακτικές το 2018, αλλά αυτό είναι ήδη αργά για να ε, ετοιμαστούν τα κράτη-μέλη και να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους για συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Ίσως λοιπόν ε, κάνουμε μια εξαίρεση στον κανόνα και διαθέσουμε δημοσίου τις πληροφορίες νωρίτερα, πριν το 2018, αλλά δεν μπορώ να προβλέψω από τώρα πότε ακριβώς ε, θα δημοσιοποιήσουμε τα σχετικά έγγραφα. Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ακαιρεότητα της Κόρσια, της αντιστάθμισης εκπομπών και προγράμματος μείωσης στη διεθνή πολιτική αεροπορία, ερώτηση Γκέρλινγκ, Λίζε, Μάισνερ, Ντάλι. Ε, ένα από τα χαρακτηριστικά της αντιστάθμισης είναι ότι στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών να μην γίνεται μόνο στον ίδιο τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας, αλλά σε προγράμματα μείωσης που γίνονται στο έδαφος και πιθανόν και από άλλους τομείς. Οπότε τα κριτήρια ε, για την αντιστάθμιση πρέπει να είναι στιβαρά και υπάρχουν κάποια κριτήρια, τέτοια στιβαρά κριτήρια στο, στις προτάσεις που θα εγκριθούν και αυτά τα κριτήρια αντικατοπτρίζουν κάποια, κάποιες περιβαλλοντικές πτυχές. Για παράδειγμα, μια εύρωστη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ε, συγκεκριμένης σημείωσης εκπομπών που επιτυχάνεται από συγκεκριμένο έργο ή σχέδιο. Για παράδειγμα, είχαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο και το μηχανισμό για τα καθαρά στήματα και εκεί ξέρουμε ε, πώς ε, μονάδες παράγονται από τη διαδικασία μείωσης. Οπότε τέτοια κριτήρια περιλαμβάνουν την προσθετικότητα, για παράδειγμα. Ένα σχέδιο, ένα έργο δεν εξασφαλίσει πληρωματικότητα, αν θα μπορούσε να είχε συμβεί και χωρίς ε, το κίνητρο της αντιστάθμισης. Κριτήρια περιλαμβάνουν και την ηχηλασιμότητα, για παράδειγμα. Τα μόρια και οι μονάδες που παράγονται θα πρέπει να ανοιχνεύονται μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης, ώστε να αποφεύγεται η διπλή καταμέτρησή τους ή η διπλή χρήση τους. Ε, η αποφυγή της διπλής καταμέτρησης είναι μία από τις αρχές που διέπουν τα κριτήρια. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κριτήρια που ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ε, περιβαλλοντική ακαιρεότητα του συστήματος Κόρσια. Επίσης, ρωτήσατε πώς ε, το θέμα των βιώσιμων καυσίνων λαμβάνεται υπόψη. Η Κόρσια προβλέπει ότι αν μια αεροπορική εταιρεία συνδυάζει βιώσιμα καύσιμα αεροπορίας στο ενεργειακό της μείγμα, οι εκπομπές της θα μειωθούν λόγω αυτής της ε, κοινή χρήσης βιοκαυσίμων και παραδοσιακών συμβατικών καυσίμων. Και αυτό είναι ένα κίνητρο για να χρησιμοποιούν περισσότερα ε, καύσιμα από ανανεώσιμε πηγές ε, στο ενεργειακό τους μείγμα οι αεροπορικές εταιρείε. Βέβαια, αυτά τα βιώσιμα καύσιμα, αυτά τα καύσιμα, τα εναλλακτικά μάλλον, θα πρέπει να είναι και βιώσιμα. Και η βιωσιμότητα είναι ένα άλλο στοιχείο της περιβαλλοντικής ακεραιότητας γιατί μας ρώτησε η κυρία Γκέρλινγκ πόσο ε, σίγουροι είμαστε ότι εξασφαλίζεται. Η περιβαλλοντική ακαιρεότητα περιλαμβάνει και το κριτήριο της υλοποίησης ενός, μιας ελάχιστης μείωσης εκπομπών αερίων του ε, θερμοκηπίου από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, τα κριτήρια περιλαμβάνουν, όπως ήταν αναμενόμενο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Δεν ε, επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στο θέμα της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ο Πίτερ Λίζε ρώτησε τι είδου ε, σχέδια και έργα εγκρίθηκαν. Στην Κόρσια δεν προβλέπονται θετικοί και αρνητική κατάλογοι για το τι είδου σχέδια επιλέγονται, είναι επιλέξιμα. Τα σχέδια πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια και μόνο τα σχέδια και προγράμματα που ε, πληρούν τα κριτήρια παράγουν ε, μόρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα της στο Κόρσια. Και φυσικά θα έχουμε και ανεξάρτητους ελεγκτές των σχεδίων και των προγραμμάτων που είναι επιλέξιμα. Το ίδιο θα ισχύσει και για την πιστοποίηση των βιώσιμων καυσίμων της αεροπορίας. Θα έχουμε δηλαδή και εκεί ανεξάρτητους επιθεωρητές. Βέβαια δεν θέλουμε επικάλυψη ό,τι αφορά τις α, ε, διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ΡΕΝΤ 2. Εδώ μιλούμε για βιώσιμα καύσιμα της αεροπορίας που χρησιμοποιούνται στη διεθνή αεροπορία. Την αεροπορία δηλαδή που δεν συμπεριλαμβάνεται σε εθνικά καθορισμένες συνεισφορές της Συμφωνίας των Παρισίων. Οπότε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κριτήρια, δεν έχουμε και καμία εγγύηση ότι τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα θα είναι και βιώσιμα. Τέλος, για να απαντήσω στην πρώτη της κυρίας Δάλη. Αν είμαστε βέβαιοι ότι η ΚΑΟ θα μειώσει τις εκπομπές της. Η ΚΑΟ γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση, γιατί ε, αναμένεται αύξηση των εκπομπών της πολιτικής αεροπορίας στο μέλλον, αλλά έχουμε μια δέσμη μέτρων, ένα σύνολο μέτρων που στόχο έχουν την την αναχέτηση της μεγάλης αύξησης ε, και μακροπρόθεσμα και τη μείωση των εκπομπών της πολιτικής αεροπορίας. Για παράδειγμα έχουμε βελτιώσει στην αποδοτικότητα ή στον, ε, έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας, ε, στην πλοήγηση και στην διαχείριση. Επίσης εναλλακτικά βιώσιμα καύσιμα, είναι ο δεύτερος πυλώνας και τρίτος πυλώνας είναι τα πρότυπα για το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή τεχνολογίες αεροναυπηγικής που χρησιμοποιούνται για να μειώνονται οι εκπομπές του κάθε τύπου αεροσκάφους. Αυτοί οι πυλώνες θα συμβάλλουν στη μείωση μακροπρόθεσμα των εκπομπών από την πολιτική αεροπορία και η Κόρση, το σύστημα αντιστάθμισης, έχει αναγνωριστεί ως σύστημα αντιστάθμισης, όχι μείωσης καθ' αυτής εκπομπής. Και ε, γεφυρώνει κάπως το κενό ε, όσο περιμένουμε πιο αποδοτικά και πιο ενεργειακά αποδοτικά αεροσκάφη και αύξηση της χρήσης των ε, εναλλακτικών καυσίμων και στην αεροπορία. Επίσης, η ΚΑΟ δεν έχει οθετήσει ποσοτικοποιημένους στόχους για τη χρήση εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων στην αεροπορία. Έγιναν συζητήσεις για το σημείο αυτό ακριβώ στο Μεξικό την περασμένη εβδομάδα και αποφασίστηκε να έχουμε αύξηση των βιώσιμων μεν καυσίμων, αλλά δεν θεσπίστηκαν ούτε καν βραχυπρόθεσμα πριν το 2025 ποσοτικοποιημένοι στόχοι. Απλώς αναφέρθηκε η ανάγκη αυξημένης χρήσης τέτοιων καυσίμων. Εγώ σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 15 της ημερησίας διατάξεως, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τον προϋπολογισμό σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων. Ο Ούγκο έχει το λόγο, παρακαλώ. Thanks uh, very much, uh, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι έλαβαν και διάβασαν την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν έχουμε πολύ χώρο ε, και ε, προετοίμασα ένα ανεπίσημο υπόμνημα ε, το και το έστειλα χτες το βράδυ. Ζητώ συγγνώμη, έχουμε πολλά σημεία ε, να συζητήσουμε. Αν θέλετε κάποιοι να συζητήσετε και να κάνετε πηγαδάκια εκτός της αιθούσης παρακαλώ εδώ έχουμε πολλά δεν με ακούνε μάλλον στην συνάδελφοι λέει ο Πρόεδρος εάν θέλετε λέω να συζητήσετε να το κάνετε εκτός της αιθούσης σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλετ παρακαλώ Έλεγα λοιπόν, Πάβο, ότι ε, προετοιμάσαμε ένα ανεπίσημο υπόμνημα όπου αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί στην στο σχέδιο γνωμοδότησης δεν έχουμε πολύ χώρο και δεν έχουμε δυνατότητα να τα αναφέρουμε όλα αναλυτικά. Γνωρίζουμε όλοι ότι ε, θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις ε, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην διαχείριση της ε, μεταναστευτική μεταναστευτικής ε, κρίσης, άμυνα στην εργασία και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, καθώς επίσης και όλα αυτά που συζητάμε εδώ, την επίτευξη των στόχων της ενέργειας που είναι φυσικά από τους πρώτους μας στόχους. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα ρεαλιστικό, ε, υλοποιήσιμο ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να ε, υλοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες και χρειαζόμαστε ένα ικανοποιητικό οικονομικό σύστημα. Θα πρέπει ένα τέτοιο σύστημα και η μεταρρύθμιση μάλλον ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρά στοιχεία αυτό που προτείνουμε ε, στην, ε, ε, στο προσχέδιό μας εδώ, στο ψήφισμά μας, είναι να είναι απτές οι αλλαγές και οπωσδήποτε να είναι ορατές στους πολίτες και να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, γιατί εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και είναι ακριβώς η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο και πρέπει πρέπει να επιτευχθούν σε ενωσιακό. Βεβαίω ε, δεν ξεκινάμε εκ του μηδενό. Ε, έχουμε και το Reflection Paper, το έγγραφο προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν τι διακοπέ και τώρα το Κοινοβούλιο ακριβώ προβληματίζεται και λέει τι απόψει του όσον αφορά ε, αυτήν την γνωμοδότηση. Ήταν η έκθεση τη κυρία Τόμα που υπερψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε και την έκθεση Μοντε που είναι ένα πάρα πολύ πυκνό πυκνό κείμενο και από το οποίο εμπνευστήκαμε. Πρόκειται για την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ε, πόρους. Όσον αφορά το περιβάλλον και τη βιώσιμη ενέργεια, ε, πολλά προγράμματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μπορούν να καταγραφούν. Ας πούμε, διασυνοριακές ενεργειακές δομές, ανάπτυξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών κλπ. Ξέρετε τα στοιχεία αυτά όλοι ε, εμείς εδώ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δεν υπάρχει λόγος να τονίσω πόσο προστιθέμενη αξία έχουν. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε να κάνω κάποιες ε, προτάσεις οι οποίες αναφέρονται ε, στο κείμενο συγκεκριμένα δηλαδή για ίδιους πόρους ε, για ενεργειακά περιβαλλοντικά προγράμματα. Ε, πρώτον το σύστημα ETS, ανταλλαγής ε, και εμπορίας ρήπων. Εγώ είμαι άλλωστε και σκιώδης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού. Θα πρέπει σύμφωνα και με την ισχύουσα ε, προ, ε, ε, την ισχύουσα διαδικασία να μοιραστούμε ακριβώς το ζήτημα, το ζήτημα αυτό. πριν από δύο χρόνια 3,6 δις, σχεδόν 4 δις ευρώ ήταν τα έσοδα από το σύστημα. Πολλά χρήματα λοιπόν και ε, υπό το νέο νομικό μεταρρυθμισμένο πλαίσιο ε, περιμένουμε ε, να έχουν αύξηση αυτά τα έσοδα για τα κράτη-μέλη. Αυτό βέβαια μας δίνει και την δυνατότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε επιπλέον ε, χρήματα τα οποία τώρα πηγαίνουν προς τις χώρες και προς τα Υπουργεία Οικονομικών των χωρών. Μας επιτρέπει λέω να προωθήσουμε, να διοχετεύσουμε τα χρήματα αυτά σε προγράμματα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που, θα μπορού, που δεν θα μπορούσαν να τα υλοποιήσουν τα κράτη μόνα τους τι λοιπόν θα ήταν μια πρώτη ενδεχόμενη ε, πηγή επιπλέον εισοδήματος. Ένα δεύτερο ε, πεδίο είναι βεβαίως οι μεταφορές και οι μεταφορές βεβαίως ε, συνδέονται με το πεδίο δράσης της δικής μας Επιτροπής. Αναφέρομαι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την καλοκαιρινή διακοπή για εναρμόνιση των ε, εθνικών ε, συστημάτων χρέωσης ε, που βασίζονται στις εκπομπές και στον, στη, στην απόσταση που καλύπτεται. Ε, βεβαίως ε, αυτό το πρόγραμμα των χρεώσεων ε, στη, για την χρήση των οδικών δικτύων θα μπορούσα να λειτουργήσουν θετικά τα προγράμματα αυτά έτσι ώστε ένα τμήμα των εσόδων να προωθηθεί για προγράμματα προστιθέμενης αξίας. Αναφέρομαι εδώ και στους αυτοκινητόδρομους, συγγνώμη, στους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, αναφέρομαι επίσης και στην εσωτερική ναυσιπλοεία κλπ. Ε, υπάρχει όμως και μία τρίτη ε, ενδεχόμενη πηγή για νέους πόρους ε, και δεν θα πω τίποτα άλλο, ε, υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία στη γνωμοδότηση αλλά δεν έχω χρόνο. Ε, ε, αναφέρομαι στην τιμολόγηση του άνθρακα. Δεν είναι το ίδιο με το σύστημα ανταλλαγής και εμπορίας ρήπων. Λοιπόν, ε, αναφέρομαι στην τιμολόγηση του άνθρακα που θα αναφέρεται στην, στο ίχνος άνθρακα ε, των ε, συναλλαγών. Ε, είχε προταθεί ένα παρόμοιο σύστημα παλιότερα, το οποίο δεν είχε γίνει δεκτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να προτείνουμε μία νέα προσέγγιση, η οποία είναι ευφυής, η οποία είναι λογική και την είδαμε και την αντιγράψαμε και στη δικιά μας έκθεση. Ε, το προστιθέμενο λοιπόν περιεχόμενο άνθρακα θα μπορούσε ε, να ε, αναφέρεται σε ποσοστό φόρου το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και θα αναφερόμαστε εδώ και στα προϊόντα γηγενός παραχθέντα και σε εισαγόμενα προϊόντα και αργότερα σε 5-10 χρόνια ένα τέτοιο σύστημα ε, θα μπορούσε ε, να συμπληρωθεί μέσω μέσω υποκατάστασης ε, τμήματος ή ολοκλήρου και του ποσοστού ΦΠΑ το οποίο αφορά πλέον, το οποίο χρησιμοποιείται για την ώρα. Λοιπόν, από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχουμε λάβει ε, και μία ε, έχουμε λάβει υπόψη μας και κάποια πρόστιμα τα οποία έχουν ληφθεί για μη συμμόρφωση προς κρατών μελών και αυτά έχουν συνυπολογιστεί τα ποσά των προστήμων και αναφέρεται άλλωστε και στην έκθεση Μόντι. Και αργότερα σε ερωτήσεις απαντήσεις μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν προτείνουμε να μπούμε ε, σε ε, διαδικασίες όπως είναι ας πούμε φόρος καυσίμων ε, ή φόρος ή δασμός για, τα, για την ηλεκτρική ενέργεια. Αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε στη γνωμοδότηση αυτή ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχει προταθεί παλιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έγινε σαφώς δεν έγινε καθόλου αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε λίγο και από το ε, παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν προτείνουμε καθόλου να ληφθούν υπόψη αυτές οι προτάσεις. Δεν είναι βέτο, αλλά αυτή την άποψη έχουμε όσον αφορά φόρο καυσίμων και ηλεκτρικού. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις προτάσεις σας. Και τώρα των πολιτικών ομάδων, η κυρία Ντάλι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή μας, τον Ιβο Μπέλετ, για την έκθεσή του. Αντικαθιστώ εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι ο σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την ομοδότηση. Ζητά συγγνώμη γιατί κολλείεται. Πάντως τον αντικαθιστώ εγώ και σας μεταφέρω το μήνυμά του. Το σύστημα το, τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ίδιων Πόρων ε, πολύ σημαντικό θέμα για συζήτηση εν ώψη το, των επικείμενων διαπραγματεύσεων και για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και για να καλυφθεί η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον κοινοτικό προϋπολογισμό μετά τον Brexit. Ευχαριστώ λοιπόν τον Ιβο για τη γνωμοδότησή του. Αποτελεί πολύ καλή βάση για συζήτηση και συμφωνώ με αρκετές προτάσεις του και θα ήθελα φυσικά να τη συζητήσουμε ε, από κοινού καθώς και τις δικές μας συστάσεις. Όντως χρειαζόμαστε σημαντικές συμπληρωματικές επενδύσεις για να ανταπεξέλθουμε στους στόχους μας που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα ήταν ε, κατά της ιδέας ενός φόρου ρηκτών καυσίμων ένας φόρος προστιθέμενο τη άνθρακα για τα, για τα διάφορα αγαθά και μια επιβολή του στα σύνορα, ώστε να αντισταθμιστεί η διαφορά μεταξύ του κόστου παραγωγής εξοκοινωτικής και ενδοκοινοτική παραγωγή. Θα καταθέσουμε μάλιστα και σχετικές τροπολογίες. Πάντω προσβλέπει ο κ. Ανδρουλάκη σε αγαστή συνεργασία και με τον Ήβο και με του υπόλοιπου και ηγητέ. Ευχαριστώ Μίριαμ. Η ΣΥΑΡ δεν έχει ορίσει ακόμη σκιώδη συγγήτη. Ε, έχουμε όμως τη σκιώδη συγγήτρια των φιλελευθέρων, την κυρία Γιάταρμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτη η συζήτηση για, την, ε, για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, Πιστεύω ότι η διπόρη θα πρέπει να είναι ε, βασική πηγή των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον. Ένας φόρος ηλεκτρικής ενέργειας ή ε, φόρος ε, καυσίμων των οχημάτων ίσως προσκρούσει σε ισχυρές πολιτικές αντιθέσεις και αντιστάσεις. Γι' αυτό δεν κρίνω σκόπιμο να προτείνουμε τέτοιους φόρους ως πηγή εσόδων για ίδιους πόρους. Επίσης, ε, σε χώρες πολύ αρεπετικημένες, ε, με πολύ μακρά δίκτυα μεταφορών ή χωρίς ε, επαρκείς υποδομές, θα είναι επιβαρυντικές οι προτάσεις. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών ε, για πολλά θέματα και οι περιβαλλοντικές προτάσεις ε, επίσης ε, θα έχουν ως αποτέλεσμα την άνηση κατανομή του κόστους μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά και περιμένουμε τη συνέχεια της συζήτησης. Thank ευχαριστώ πολύ. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ να κλείσετε το μικρόφωνο σα. Σα <laughs> ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η επόμενη ομιλητρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω δύο-τρία λόγια. Να ευχαριστήσω καταρχά ε, τον συνάδελφο, τον κύριο Μπελέτ, που προετοίμασε το κείμενο αυτό. Σε ό,τι αφορά το μέλλον τώρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση και το παρελθόν. Να μάθουμε, να διδαχθούμε το παρελθόν, να προσπαθούμε να έχουμε υπόψη μας κατά πόσον μπορούμε πραγματικά και αποτελεσματικά να χρησιμοποιούμε τις ήδη φυστάμενους πόρους, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε ακόμα δυσκολίε σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική θέση των εφιστάμενων πόρων. Ας μην επαναλάβουμε και στο μέλλον τα ίδια λάθη. γιατί κάποια κρατημέλη εξακολουθούν να προστατεύουν τις αγορές τους. Ακόμα και αν δεν πρέπει να το κάνουν και αντί να χρησιμοποιούν πιο πολύ ηλεκτρισμό από τον άνθρακα, ενώ δεν θα έπρεπε και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τι θα κάνουμε στο μέλλον αν ήδη σήμερα δεν πληρούνται κάποιοι όροι. Κοιτώντας τώρα το μέλλον, Υποστηρίζουμε προφανώς ε, πιο συγκεκριμένα project και έργα θα θέλαμε και earmarking ορισμένων πόρων για τέτοιους σκοπούς. Από την άλλη, καλωσορίζουμε τη δήλωση του εισηγητή ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο πολλά συστήματα τύπου ETS, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και να εφαρμόσουμε πιο πολλούς φόρους για την χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων. Να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να μην προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε πολλά και διαφορετικά. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή πολιτική σε διάφορες περιστάσεις και θα θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τα όσα λέει και ο εισηγητής. Ωστόσο, έχω κάποιες ανησυχίες για ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε στην έκθεση βασικά. Στην παρούσα φάση κάποια κρατημέλη χρησιμοποιούν ήδη έσοδα από το ETS για πράσινα προγράμματα και έργα. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι στην τελική ανάλυση τα κράτη αυτά δεν θα χάσουν πόρους στο μέλλον, γιατί κάποιες χώρες ήδη στην παρούσα φάση παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεν θέλουμε να τιμωρηθούν ουσιαστικά αυτές οι χώρες στο μέλλον επειδή ήδη δραστηριοποιήθηκαν πιο νωρίς από ό,τι άλλοι. Δεν θέλουμε να του αφαιρέσουμε δηλαδή κάτι το οποίο ήδη κάνουν. Ασφαλώς και είναι πάρα πολύ θετικό και συμβάλλει πολύ στην ευημερία των, Ευρωπα... των Ευρωπαίων πολιτών. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε και προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία. Να πω επίση ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερω που η Επιτροπή μα. Ε, εργάζονται επί τη έκθεση αυτέ. Δεν θα πρέπει να παραμείνει αυτό μόνο στο πεδίο εφαρμογή τη επιτροπή Ελέγχου του Επιτροπή Προπολογισμού. Ο κύριο Eichhout. Κύριε Eichhout, είστε εδώ στην αίθουσα παρακαλώ. Όχι. Δυστυχώ αποχώρησε. Μάλιστα. Η ευθυντή τώρα. Ο κύριο Πελιτσίνη. Ούτε αυτό. Η ΕΝΕΦ. Πολύ ωραία. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μοντανιόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τη δυνατότητα ε, να δώσω και εγώ κάποια στοιχεία όσον αφορά αυτό το θέμα, επί του οποίου αναφέρθηκε ο εισηγητής σε αδρές γραμμές. Ε, να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία, πρόκειται για ένα θέμα πολύ δύσκολο. Ε, πρέπει να ψηφιστεί με ομοφωνία, χρειαζόμαστε επικύρωση επίσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια και εδώ και 30 χρόνια προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ε, και ε, συστηματικά οι διαπραγματεύσεις ε, αποτυγχάνουν με την έγκριση του προηγούμενου ε, πολιετούς ε, πλαισίου έγινε μια προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση αυτή και δημιουργήθηκε λοιπόν η ομάδα Μόντι με τρεις Ευρωπαίους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τρεις επίσης επιτρόπους και εκπροσώπους του Συμβουλίου που προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα αυτό. Προσπαθήσαμε λοιπόν έτσι ώστε να, συλλέξουμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε ρυθμίσουμε την επόμενη φορά το σύστημα. Όπως είπατε θα πρέπει να ξαναδούμε ε, το σύνολο του προϋπολογισμού. Και εδώ ακριβώς η έννοια της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναλαμβάνει πλέον ε, όλη την σημασία των όρων γιατί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, δεν είχε πάντα ε, σχέση με την προστιθέμενη αξία, αλλά η έννοια της, η έννοια των ίδιων πόρων είναι ότι και από την πλευρά των δαπανών να βρούμε μια προστιθέμενη αξία. Όταν λοιπόν ορίστηκαν οι υποψήφοι, επί των οποίων εργάζεται η Κομισιόν. Ε, έχουμε και ε, τα ενδεχόμενα green basket όσον αφορά τις μεταφορές και το περιβάλλον ας πούμε και γι' αυτό λοιπόν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για την, Επιτροπή, για την έκθεση Επιτροπής Προϋπολογισμού προς ώρας σκεφτόμαστε δεν έχουμε για την ώρα αποφασίσει, δεν έχουμε προσθέσει κάτι, δεν έχουμε αφαιρέσει κάτι. Ε, ε, στην διάλεξη για την ε, κατάσταση της ενώσεως και στην ομιλία της Ορβόνης έχουν αναφερθεί κάποια στοιχεία σχετικά με το θέμα. Υπάρχει ο έλεγχος των συνόρων που ίσως διευρύνθηκε περισσότερο από λόγω καταστάσεων συγκεκριμένων. Εν πάση περιπτώσει, ε, η Κομισιόν ακόμα ε, δεν έχει πάρει αποφάσεις. Τον Μάιο του 2018 θα υποβάλει προτάσεις, ε, όταν δηλαδή θα κάνει τις προτάσεις της και για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί και τα έσοδα εκεί εντάσσονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος. Τώρα τελικά σχόλια από τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πάβελ, και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις πολύ επικοδομητικές τους ε, παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές ε, συγκλίνουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια εκκρεμή θέματα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω, αλλά πιστεύω ότι γενικώ ε, είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος. Η κυρία Ντάλη είπε μέσα του κυρίου ε, μάλλον και ο Σαντράκης μέσω της κυρίας ε, Ντάλη, το σημείο 9 ε, και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα του φόρου θέμενο άνθρακα. Επίσης η κυρία Γιατενμάκη ε, είπε και το σημείωσα για τα πιθανά προβλήματα που θα έχει η χρέωση της χρήσης του δικού δικτύου, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν μεγάλη έκταση οδικού δικτύου. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε από υπάρχουσες εθνικές εισφορές και φόρους που ήδη εφαρμόζονται και μετά θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ίσως μια προσημείωση των κονδυλίων αυτών στο μέλλον. Η κυρία Γιατανμάκη είπε ότι δύσκολο θα ήταν, για να μην πούμε αδύνατο, να εφαρμόσουμε φόρο ηλεκτρικής ενέργειας ή τέλος καυσίμων αυτοκινήτων σε κάποια οδικά δίκτυα χώρων μελών. Θα το εξετάσουμε. Πάντως συμφωνώ και εγώ ότι δεν έχει οριμάσει αυτό το θέμα. Η κυρία Κονέτσνα μίλησε ιδιαίτερα για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Συμμετέχουμε και οι δύο στις διαπραγματεύσεις και συμφωνούμε. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη, το τι κάναμε στο παρελθόν, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους. Σε ό,τι αφορά πάντως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε την πεπατημένη και να έχουμε διαθέσιμο σύστημα, να μην σπαζοκεφαλιάζουμε, να δημιουργούμε νέα συστήματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να ε, τιμωρούμε τα κράτη-μέλη για ήδη λιμένες προσπάθειες ε, Εννοείται αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε ε, το σύστημα και ίσως να έχουμε συμπληρωματικές προσημειώσεις εσόδων από το ETS και ίσως ε, να, αντίστοιχα να μειωθούν ε, οι συνεισφορές που, ε, που απορρέουν από το καθάριστο εγχώριο εισόδημα. Σωστά το επισήμανε η κυρία Κονέτσνα. Ε, πάντως θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε η κυρία Μοντανιά και φυσικά και με τους και ηγητές ε, όσο προχωρούμε στις συζητήσει τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα, ευχαριστώ. 27 Οκτωβρίου 2017, 11 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε το Δεκέμβριο 7 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή, 22 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην Ολομέλεια το Μάρτιο του 2018. Επόμενο σημείο τη τη διάταξη είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την προαγωγή των πρωτεϊνικών καλλιεργειών ε, και ε, κίνητρα για την παραγωγή πρωτεϊνούχων και ψυχαθών φυτών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Χελβένη Γεώργη είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Είμαι πανευτυχής που έχω τέτοια δυνατότητα σήμερα. Θα ήθελα να επισημάνω ένα πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια και είναι ακόμη ανεπίλητο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από έξι χρόνια υιοθέτησε ένα παρόμοιο ψήφισμα στο οποίο επισημέναμε την ανάγκη ε, της των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι δυστυχώς μόνο 3 με 4% του συνόλου των ε, αρρώσιμων καλλιεργιών. Πολύ χαμηλό ποσοστό λοιπόν των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών και το επισημάνουμε ήδη στο ψήφισμά μας του παρελθόντος. Ενώ ε, το 70% των πρωτεϊνών που χρειαζόμαστε οφείλουμε να το εισάγουμε δεν καταφέρουμε να παράγουμε πρωτεΐνες για να ε, είμαστε αυτάρκεις. Εισάγουμε τις πρωτεΐνες μας κυρίως από τη Βόρεια Αμερική και κυρίως πρόκειται για γενετικώ τροποποιημένη σόγια και ελαιοκράβη. Οι στατιστικές όμως των τελευταίων χρόνων καθιστούν σαφέστατη και επιτακτική την ανάγκη μιας πιο συνολικής στρατηγικής πρόθεσης των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ε, πόρους μας και να αντισταθμίσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγωγές πρωτεϊνούχων καλλιεργιών, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν πρωτεΐνες που δεν θα είναι ε, γενετικά τροποποιημένες, θέλουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και γι' αυτό και δίνουμε μάχη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τη γεωργία μας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, προκειμένου να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις αγωγές και να διασφαλίσουμε μια ε, γεωργία χωρίς γενετικώς ε, τροποποιημένους οργανισμούς. Πάντως χαίρομαι που το 2013 ήδη η Ουγγαρία υιοθέτησε τη δική της στρατηγική για την προώθηση πρωτοενοχών καλλιεργειών και μάλιστα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για πρωτεΐνη απαλλαγμένη από γενετικώς στραπαπημένους οργα... οργανισμούς. Και μάλιστα χαίρομαι για την υιοθέτηση και των προδιαγραφών ε, για τη σόγια του Δούναβη και την Ευρωπαϊκή Σόγια. Επίσης είχαμε τον Ιούλιο μια γερμανογκρική πρωτοβουλία και 18 χώρες μέλη προσυπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη της Σόγιας που στόχο έχει τη διαφύλαξη της βιώσιμης γεωρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών, ιδιαίτερα μη, μη γενετικώς τροποποιημένης σόγιας. Το σχέδιο α, γνωμοδότησής μου επικεντρώνεται στις εξής προτάσεις. Ε, πρόκειται για γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Γεωργίας που είναι αρμόδια κατ' ουσία. Οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην Ευρώπη εξυπηρετούν το στόχο της ε, αηφόρου γεωργίας, ε, βελτιώνει το αποτύπωμα άνθρακα και συμβάλλει σε πιο διαφοροποιημένα αγροοικολογικά συστήματα. Επίσης μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τεχνητών λιπασμάτων με, την, με τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που είναι άζωτο και άρα μειώνουν την ανάγκη χρήσης ε, αζωτούχων λιπασμάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας ε, στην καινοτομία και στην τεχνολογική έρευνα. Οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ε, και τα ψυχανθή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα ψυχανθή δεν προορίζονται μόνο για ζωοτροφές. Επίσης, θέλουμε ε, μια πιο ανταγωνιστική παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα έχουμε να υποστούμε τον ανταγωνισμό των προϊόντων από τρίτες χώρες. Αυτά σε γενικές γραμμές ε, λέω στην γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τώρα οι εισηγητές, σοσιαλιστές και δημοκρατές πρώτοι. Ο κύριος Φόλκαν που αμαν... αντικαθιστά την κυρία Μελιόρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εκπρόσωπο την κυρία Μέλιορ, την σκιώδη γητρία, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Καλώς ορίζει το σχέδιο της γνωμοδότησης του συναδέλφου η κυρία Μέλιορ και συμφωνεί σε μεγάλο ποσοστό. Έχει κάποιες μικρές αλλαγές να προτείνει στο κείμενο. Ένα σημείο το οποίο ε, δεν συμφωνεί απόλυτα είναι στο σημείο 7 για τη νέα αξιολόγηση για την απαγόρευση των παραστακτών σε κάποιες οικολογικές εκτάσεις. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να επηρεάσει πάρα πολύ τη βιολογική βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυρία Μέλιορ θεωρεί ότι η προτινόμενη νέα αξιολόγηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόμενη άρση της απαγόρευσης που έχει πολύ θετικέ επιπτώσει. Αυτά εν συντομία σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση και την τοποθέτηση τη κυρία Μέλιορ. Προσβλέπει στη μελλοντική συνεργασία και εύχεται κάθε επιτυχία στι μελλοντικέ εργασίε. Ευχαριστώ και εγώ. Από το ECR τώρα, ο κύριος Ντόρμαν. Δεν είναι στην αίθουσα. Από την άλλη, λοιπόν, η σκιώδηση, η κυρία Γιατεμάκη. Ευχαριστώ, πρόεδρε, συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έκανε εξαιρετική σύνοψη των όσων συμβαίνουν και των όσων διακυβεύονται στην παρούσα φάση. Η παραγωγή πιο πολλής πρωτενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει πολλά ωφέλη, πραγματικά και σημαντικά ωφέλη. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρω την ευκαιρία αυτή που έχουμε στη διάθεσή μα αυτή τη στιγμή. Η έλλειψη των πρωτενούχων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γεγονό. Εισαγάγουμε 70 περίπου των αναγκών μας. Μειώνοντας λοιπόν τις εξαρτησή μας από τις εισαγωγές θα έχουμε πιο πολλά μέσα και εργαλεία στα χέρια μας. Θα μπορέσουμε να μειώσουμε την πίεση σε πολύ ευάλωτα οικοσυστήματα εκτός Ευρώπης και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και την, το γεωργικό κλάδο να καταστεί πιο βιώσιμος. Αυτό θα είχε θετικές επιπτώσεις τόσο και στο γεωργικό εισόδημα όσο και στην βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μακρύς ο δρόμος για μια πιο βιώσιμη τέτοια καλλιεργία ενούχων. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα, το κόστος το οποίο είναι πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την παραγωγή σε σχέση με την εισαγωγή. Άρα θα έχουμε δυσκολίες για να ανταγωνιστούμε φτηνές τροπικές εισαγωγές. Ωστόσο, αν θέλουμε να κοιτάξουμε το μέλλον και να είμαστε και συνεχτικοί σε ό,τι αφορά την νομοθεσία μας ε, για την βιωσιμότητα διαφορών κλάδων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλη την ε, εικόνα, το σύνολο της εικόνας ε, και όχι τις λεπτομέρειες. Η επιτυχία για την ε, παραγωγή, το εισόδημα για τους αγρότες και η καθαρή συνείδηση. Όλα αυτά προαπαιτούν ε, ισχυρή δράση και θα ήθελα να ζητήσω μάλιστα και μια Ευρωπαϊκή Ένωση Πρωτεϊνών. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τον ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Πρόεδρος, την κυρία Γετεμάκη. Επόμενος κοιότης από την ΚΟΕ, ο κύριος Φλάναγκαν. Τον αντικαθιστά κανείς? Όχι. Να συνεχίσουμε λοιπόν ε, με τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου Μάρτιν Χάουζιν και ζητά συγγνώμη για την ε, απουσία. Ο Μάρτιν είναι ο υπεύθυνος αλλά ε, αυτό που φοβάται είναι ότι ενδεχομένως ε, αυτή η διάταξη θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί η εισαγωγή ε, γενετικώς τροποποιημένης σόγιας οι προκλήσεις ε, της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλες ε, και βλέπουμε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να προωθηθεί στην Ευρώπη η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων ε, καλλιεργειών αλλά μη γενετικώς τροποποιημένων ε, το ζήτημα είναι το κατά πόσον ε, οι, ε, οι οικολογικές περιφέρειες τελικά θα ενθαρρύνουν, θα ενθαρρυνθούν για την καλλιέργεια μη γενετικώς τροποποιημένων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και όχι να έχουν στόχο μόνο την αύξηση της παραγωγής. Επίσης θα πρέπει να γίνει λόγος και για τη μείωση των, ε, των εντομοκτώνων. Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί ενδεχομένως ως βιώσιμη και η καλλιέργεια για ε, την ε, παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως πούμε η ελαιοκράμβη. Επίσης ε, υπάρχουν ε, στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ενώ ε, προωθείται, υποτίθεται η μη γενετικώς τροποποιημένη σόγια σε πολλές ή οποιαδήποτε άλλη πρωτεϊνική καλλιέργεια, το γεγονός της εντατικής μονοκαλλιέργειας τελικά δίνει αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να προωθηθεί η, ε, ε, η καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων ε, σε γη στην οποία επιτρέπεται να βοσκήσουν και τα ζώα γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο βιώσιμη η καλλιέργεια. Επίσης, να πω το εξής, κάτι που δεν ανέφερε κανείς. Εάν πάρεις κανείς την πρωτεΐνη του από από, την, ε, από φυτικές παραγωγές, ε, τότε κερδίζουμε ε, και τις πρωτεΐνες, τις οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να πάρουμε από το κρέας, γνωρίζοντας τις συνέπειες που αυτό, αυτό που έχει και είναι ένα σημείο το οποίο δεν ανέφερε κανείς από τους προλαλήσαντες. Επομένως, ναι, εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εμείς ε, ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την εργασία που έχει κάνει και εμείς με τη σειρά μας αναγνωρίζουμε ε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό και για τους καταναλωτές και για τους γεωργούς. Επίσης θετικά τα αποτελέσματα και για το περιβάλλον και για τη μείωση του αζότου στην ατμόσφαιρα των εκπομπών, σημασία για το περιβάλλον και σημασία επίσης και όσον αφορά τις ζωοτροφές. Ε, να σας πω, σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, ε, υπάρχει μία μακρά παράδοση με καλλιέργεια λούπινου, φουλιού κτλ ε, για την κυρίως για χρήση σε ζωοτροφές ε, και πιστεύουμε ότι αυτές ε, οι παραδόσεις μας πρέπει να διατηρηθούν. Αυτή τη στιγμή τώρα το 70% των ζωοτροφών καλύπτεται από εισαγωγές και όλες οι ζωοτροφές, οι περισσότερες τουλάχιστον έχουν βάση τη σόγια η οποία είναι και γενετικώς τροποποιημένη και επομένως η ε, ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος με τις δικές μας ε, παραγωγές. Ε, επίσης στις αρρώσιμες γεές χρησιμοποιούνται ουσίες εντομοκτώνα, ζυζανιοκτώνα και ένα σωρό άλλα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στις καλλιέργειες. Εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα ε, στο θέμα της, ε, στα πλαίσια μάλλον της ε, αναθεώρησης της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε μια και μιλάμε για προστατευόμενες καλλιέργειες. Σας ευχαριστώ κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ χαιρετίζω αυτήν τη στρατηγική ε, για τα πρωτεϊνούχα, κυρίως γιατί και εμείς στη Γερμανία, στην Βαβαρία αλλά και στην Αυστρία έχουμε ήδη εγκρίνει ε, την στρατηγική της εσόγες του Δούναβη και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι πολλά στοιχεία από αυτή τη στρατηγική αναφέρονται και εδώ. Το σημείο 7 ε, είναι, της έκθεσης για μένα είναι ε, σημαντικό. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να ξαναδούμε ε, τι αναφέρεται σχετικά με τις επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος. Εδώ ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 300.000 εκτάρια τα οποία προστατεύονται ε, ε, εννοώ προστατεύεται η βιοποικιλοτητα τους και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και άζωτο το οποίο αποθηκεύεται στις περιοχές αυτές και βεβαίως εάν ένας γεωργός αποφασίσει να καλλιεργήσει σιτάρι ή κάποια άλλα σιτηρά ξέρουμε ότι ε, θα είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι τα πρωτεϊνούχα και φυτά και επομένως θα πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια πειθούς των γεωργών. Πρέπει επίσης ε, να πούμε ότι ναι να διατηρηθούν ε, και τα πάρκα και οι πράσινοι χώροι χωρίς όμως να να λησμονούμε και τα λιβάδια, γιατί ε, ε, στα λιβάδια θα πρέπει να τρέφονται τα ζώα μας. Σε γενικές γραμμές ε, μπορώ να πω ότι εκτιμούμε θετικά αυτήν την πρόταση. Κύριε Ντάλη, ευχαριστώ. Όντω το θέμα είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντική στρατηγική πρωτεΐνοχων καλλιεργιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η σημασία των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών φάνηκε και στα πλαίσια της συζήτησης για τα βιοκαύσιμα και τις οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι συναφές ε, και με την εξάρτησή μας ε, από τις εισαγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Και γι' αυτό ε, με την αύξηση της παραγωγής σόγιας και την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών σε ευρωπαϊκές χώρες θεωρώ ότι θα έχουμε ένα ευρύ φάσμα πλέον εκτιμάτων και ταυτόχρονα θα μειώσουμε τον άζωτο στην ατμόσφαιρα, θα χρησιμοποιούμε λιγότερα λιπάσματα που γίνονται με βάση ορυκτά καύσιμα, θα μειώσουμε τις, τα επίπεδα ασθενειών, θα προστατεύουμε τη βιοπικιλότητα και θα ενισχύουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή ζωοτροφών, μειώνοντα την εξάρτησή μα και θα το συνδυάζουμε αυτό με την τρέχουσα συζήτηση για τα βιοκαύσιμα. Θα είναι θετική η επίπτωση ε, και για τους γεωργούς. Ε, θα αυξάνεται το δυναμικό πρωτενούχων καλλιεργιών ε, δυνάμει της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και με τη στρατηγική αυτή μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να καλλιεργούν μη γενετικώς τροποποιημένες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει η κυρία Μούλκερ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα κάνω ε, μία σύντομη αναφορά στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ε, των διατάξεων που αφορούν τη γεωργία από τον κανονισμό Omnibus. Στις 12 Οκτωβρίου έχουμε καταλήξει συμφωνία και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει και επιβεβαιώνει την πρόθεσή τη να αναθεωρήσει την κατάσταση προσφοράς και ζήτησης πρωτεΐνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική πρωτεϊνούχων καλλιεργιών. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε τις εσωτερικές προετοιμασίε, την εξέταση του πεδίου εφαρμογή και τα στοιχεία ενό τέτοιου ευρωπαϊκού σχεδίου πρόθεσης των πρωτεϊνούχων καλλιεργιών σε στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενους και φυσικά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένουμε χαιρετίζοντας την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας για το θέμα αυτό προκειμένου στο μέτρο του δυνατού να ευθυγραμμιστούμε ε, στην, ε, στις ιδέες και την υποβολή του σχεδίου με τις προτάσεις Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Επαναρχόμαστε στον εισηγητή μας τον κύριο Χολβένη για τα τελευταία σχόλια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Τι σημείωσα, θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη. Ευχαριστώ καταρχήν για την υποστήριξή σας. Και είναι σαφές ότι κάποια σημεία θα θα τα συζητήσουμε διεξοδικότερα, το θέμα των βιοκαυσίμων και το θέμα των φυτοφαρμάκων. Δεν πρόκειται να επισέλθω εδώ σε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως, ε, όντως, ε, και αυτά τα δύο θέματα είναι συναφή και κέρια και για το αντικείμενο που μας απασχολεί. Ευχαριστώ και πάλι. Ωραία, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή. Μην ξεχνάτε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που λήγει στις 27 Οκτωβρίου στις 11 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 7 Δεκεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τον ορισμό παρουσίαση και επισήμαση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμαση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της έκθεσης ε, Αγιούσο και θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Πιλάρα Αγιούσο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κάναμε πολλές ε, ε, συναντήσεις και να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής μας εδώ καθώς επίσης και τη γραμματεία της ομάδας μου γιατί δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ για αυτήν την ε, έκθεση. Γνωρίζετε ότι η ψηφοφορία προτείνεται, ε, προβλέπεται συγγνώμη, για τις 28 Νοεμβρίου και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και την πρώτη συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές. Επομένω, σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε τα διάφορα ε, σχόλια από πλευρά των βουλευτών, όσων τουλάχιστον ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, ε, σχόλια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα τις συμβαστικές τροπολογίες. Έχουν υποβληθεί πολλές ε, ε, τροπολογίες, 44 από την πλευρά διεθνής, διεθνούς εμπορίου. Έχουμε και τροπολογίες από πλευρά της Επιτροπής Γεωργίας που δεν έχουμε στη διάθεσή μας λόγω των τεχνικών προβλημάτων που είχαμε ε, αυτή την ε, εβδομάδα. Επίσης, ε, επί των παραρτημάτων σίγουρα υπάρχουν πολλές τροπολογίες, οι οποίες οπωσδήποτε θα είναι στη διάθεσή μας. Τώρα έχουμε τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ τη Γραμματεία που έχουν κάνει τα πάντα έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις τροπολογίες αυτές. Επίσης, παρακαλώ να παρακαλώ Στου του συναδέλφους να μελετήσουν προσεκτικά τι τροπολογίε του να δουν αν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων όσον αφορά ε, το θέμα της διευκρίνησης ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Πιστεύω ότι την πρόταση ε, αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να την ευθυγραμμίσουμε με όσε πολιτικές τροποποίησει έχουν προέλθει λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίε όσον αφορά το θέμα αυτό και το θέμα των αρμοδιοτήτων και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική πράξη ε, έτσι ώστε να τροποποιηθεί ε, το κείμενο αναλόγω. Συμφωνώ απολύτως με τις τροπολογίε που έχουν υποβληθεί με στόχο την ε, διευκρίνηση του θέματος ότι, ε, ε, που αναφέρονται μάλλον στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και που θα πρέπει να ισχύουν και για προϊόντα τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ζητώ από την Επιτροπή λοιπόν να διευκρινίσει και νομοθετικά κάποια ζητήματα επί των οποίων υπήρξε ομοφωνία και στις τρεις αρμόδιες συναρμόδιες επιτροπές. Ε, επίσης, στην ισχύουσα νομοθεσία ε, υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται η προσθήκη ε, ενδείξης στην γλώσσα της περιοχής σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποτελεί νομική υποχρέωση στην εν λόγω περιοχή ή χώρα. Ε, το άρθρο 4 της ισχύουσας ε, νομοθεσίας ε, θεωρώ ότι παρουσιάζει ένα πρόβλημα και η Κομισιόν λέει ότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψει πρόβλημα εάν αναφερόμαστε σε γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό έτσι ώστε να πληροφορηθούν καταλήλως όλοι οι συνάδελφοι. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση γιατί δεν είναι αρκετά σαφής η Κομισιόν. Να μας το ξεκαθαρίσει λοιπόν. Έχουν υποβληθεί επίσης τροπολογίες ε, ε, που αφορούν την ε, διαφοροποίηση γεωγραφικών ενδείξεων και προστατευμένων ονομάτων μη καταγεγρεμένων. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει γεωγραφική ένδειξη όσον αφορά το κρασί ή όσον αφορά άλλα προϊόντα και τι σημαίνει μη καταχωρημένη ιστορικά αποδεδειγμένη όμως ένδειξη Επίσης, ε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει ε, η το, το αλκοόλ, ε, το ινόπνευμα θα πρέπει να είναι ε, προέλευσης ε, φυτικής βεβαίως, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που λένε ή από προερχόμενα στοιχεία από την μπύρα. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης, ενδεχομένως υπάρχει κάποιος λόγος που έχει προσθεθεί, γιατί και η ίδια η μπύρα έχει προέρχεται από ε, ενόπνευμα, από φυτική προέλευση. Επίσης υπάρχουν και κάποια στοιχεία τεχνικής φύσεως. Ε, κατανοώ βεβαίως ότι υπάρχουν προβλήματα και μένα με προβληματίζουν θέματα τα οποία άπτονται της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, αλλά δεν είναι το σωστό πλαίσιο αυτός ο κανονισμός έτσι ώστε να συζητηθούν, να αναφερθούν τα στοιχεία αυτά, άρα δεν μπορούν να γίνουν ε, αποδεκτά στοιχεία τα οποία αφορούν και τη στρατηγία του ενόπνευμα γενικά κλπ. Πιστεύω ότι οι τροπολογίε οι οποίε έχουν υποβληθεί αποτελούν μια ικανοποιητική βάση για να αναπτύξω την πρότασή μου. Βεβαίω σα επαναλαμβάνω ότι είμαι στη διάθεση όλων για προτάσει κλπ. Και, και βεβαίω ε, θέλω εδώ να σα ακούσω όλου προσεκτικά έτσι ώστε να ε, λάβω υπόψη τα στοιχεία αυτά για, την, ε, για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να ακούσουμε κάποιους ε, αντικαταστάτες ε, των σκιωδών για τους σοσιαλιστές, ο κ. Γουλκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εκ νέου ε, τη συνάδελφο κυρία Μίλια που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Με μεγάλη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον άκουσε η κυρία Μελία τη συζήτηση αυτή. Διάβασα και τι 500 και πλέον τροπολογίε. Μερικέ εξ αυτών τι κατέθεσε και η ίδια. Και η συνάδελφο είναι πολύ αισιόδοξη σε ό,τι αφορά τι επόμενε συναντήσει των σκιονδών. Θεωρεί ότι για τα πιο πολλά σημεία θα υπάρξει συνένεση και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά τον τρέχοντα κανονισμό, η ουσία είναι η μία, η καλύτερη ποιότητα των αλκοολούχων στην Ευρώπη και επί τριών σημείων θα ήθελα να εκφράσω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις από πλευρά της κυρίας Μέλια για θέματα τα οποία έθιξε άλλωστε και η συγγήτρια. Η πιο δύσκολη συζήτηση η οποία θα γίνει είναι μια συζήτηση μάλλον τεχνικής φύσεως παρά το γεγονός ότι τα πιο πολλά είναι ο πνευματώδη εδώ και πολύ καιρό εντάσσονται στα πλαίσια μιας διαδικασίας. Ε, πάντα χρειάζεται ανανέωση και μεταξέλιξη των συστημάτων. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις θα πρέπει να αποτυπωθούν και στον κανονισμό για τα ενοπνευματώδη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμπεριελήφθηκε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ακόμα να το διευκρινίσουμε. το ερώτημα είναι κατά πόσον θα γίνει αυτό μέσω εφαρμοστική ε, πράξη ή πράξη κατά εξουσιοδότηση ή μια κανονική ε, μιας κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Η κυρία Μέλια κλείνει προς την τελευταία ε, λύση, προς την κανονική νομοθετική διαδικασία. Η παραγωγή αλκοολούχων έχει μια μακρά παράδοση και σε ό,τι αφορά τον την προσαρμογή των όρων και των ορισμών. Αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει ο ορισμός των αλκοολούχων να θεωρηθεί πυρήνα όλου του νομοθετήματος. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στους ορισμούς χωρίς ε, έγκριση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Προτείνεται λοιπόν από πλευρά τη κυρία Μέλια η κανονική νομοθετική διαδικασία. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη χρήση ζάχαρη στα ανεπνευματόδη, η κυρία Μέλια θα ήθελε για κάποια ανεπνευματόδη να περιορίζεται η επιτρεπόμενο όριο χρήση ε, ζάχαρη από πλευρά των παραγωγών σε ό,τι αφορά την επιρροή της γεύσης μέσω ζάχαρης. Αυτό είναι κάτι το οποίο η κυρία Μέλια το δέχεται, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει η κατάχρηση της ε, ποσότητας ζάχαρης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την, τα τόδι από δημητριακά προτείνει καταναλωτόριο 10 γραμμάρια στις τροπολογίες της. Τελευταίο σημείο, σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δέχεται αυτό η κυρία Μέλια. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίζεται ότι οι προστατευόμενες ενδείξεις που ως τώρα ήταν στο σημείο τρία του κανονισμού να εξακολουθήσουν να ισχύουν και η κυρία Μέλια θεωρεί ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και για τους καταναλωτές αλλά και για τους παραγωγούς, για το νέο μητριό στο διαδίκτυο, το νέο online ε, μητριό θα πρέπει και αυτό να υποστηριχθεί και να δημορφωθεί σωστά έχει καταθέσει τροπολογίες. Θα υπάρξει συνάντηση των σκιωδών στο Στρασβούργο και είναι αισιόδοξο για την εξέβρεση συνένεση εσύ, κυρία Μέλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάθιος, ο οποίος αντικαθιστά την Πέτρη. Ah. <laughs> Thank you, Chairman, and thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά που έκανε στο θέμα αυτό και να πω δύο λόγια εξ ονόματος του συναδέλφου μου. Η ομάδα του ECR έκανε κάποιες τεχνικές προσαρμογές στο σχέδιο κανονισμού για να προωθηθούν και να συνεχιστούν στοιχεία από τον παλιό κανονισμό, να προστατευτούν τρόποι παραγωγής και να μην είναι υπερβολικά επαχθείς οι κανόνες για την παραγωγή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια βασικά σημεία της τοποθέτησής μας σε ό,τι αφορά και τις απόψεις της Επιτροπής. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι τα ενοπνεύματόδη θα πρέπει να θεωρείται προϊόν της ε, του τόπου παραγωγής. Και αυτό για τον χώρο που πραγματικά ε, έγινε η παραγωγή, όχι εκεί που έγινε η βασική μεταποίηση, σε ό,τι αφορά τα μείγματα, σε ό,τι αφορά και τη γεωγραφική ένδειξη, ενδεχομένως να μην μπορούν να ζητήσουν τη χρήση τη γεωγραφική ένδειξη παρά τι ε, ισχυρού παραδοσιακού ιστορικού δεσμού, Κατά δεύτερον, έχουμε κάποιε ανησυχίε ότι αφορά τη μετάφραση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όταν ένα πραγματάτης εξαγάγεται θα πρέπει να έχει ε, ετικέτα εύκολα κατανοητή για τον ε, την αγορά ορισμού. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυσκολεύει τα πράγματα και μόνο νομοθετικές πράξεις σε κάποιες καταξαίρεση περιπτώσεις. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που είχαμε τα 15, χρόνια, τα 15 τελευταία χρόνια στον τομέα των πνευματοδών, ακριβώ τέτοιου είδου περιορισμού θα πρέπει να καταργήσουμε. Θέλουμε μια απλή προσέγγιση, όπω αυτή του 110 του 008, που προτείνει ένα απλό τρόπο για τη μετάφραση για τις εξαγωγές. Κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, να υπάρχει μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας, να μπορεί να παρέμβουν οι αρχές σε, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο θέμα με την ετικέτα. Περιπιστεύουμε ότι η νέα αγορά δεν κάνει αρκετά για να προστατεύει από απάτες τους παραγωγούς και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να καταθέσουμε μια τροπολογία για να υπάρχει τέτοια προστασία των ε, βέλτιστων αυτών προτύπων σε ό,τι αφορά και την ε, σχετικό κανονισμό. Περσινές μελέτες καταδεικνύουν ότι πάνω από 4% ε, των ανεπνευματοδών χάνονται σε ό,τι αφορά πωλήσει απατηλών ενώθων προϊόντων. Πιστεύουμε ότι και στις περιπτώσεις που εισαγάγονται ενώθα προϊόντα στην Ένωση χωρί έγκριση και τέλο, υποστηρίζουμε τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, δεν πιστεύουμε αρμόνιση ότι θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό. Ο κλάδο των υμνοπνευματοδών έχει πολλέ ιδιαιτερότητε. Δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό με τι εμπειρίε από άλλου τομεί. Θέλουμε λοιπόν να τα δείξουμε τα θέματα αυτά τι επόμενε εβδομάδε στα πλαίσια τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρο. Η κυρία Μιούλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για την δουλειά που έχει κάνει ήδη ο κανονισμός για τα είναι πνευματόδη αποτελεί ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα και νομικό πλαίσιο. Από πλευρά των καταναλωτών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα είναι πνευματόδη είναι υψηλή ποιότητα και ότι τελικά ο καταναλωτή παίρνει και αγοράζει το προϊόν το οποίο περιμένει λόγω τη ετικέτα. Από πλευρά τη βιομηχανία του οικονομικού κλάδου θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφέ νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι και εύρυθμο. Αυτό αφορά και το σύστημα της γεωγραφικής ένδειξης που ε, θεωρείται και θα πρέπει να θεωρείται ως παράλληλο του συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων στο ό,τι τρόφιμα. Ο διάβολος κρύβεται συνήθως στις λεπτομέρειες, γι' αυτό χαίρομαι για τις προτάσεις που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Οι τροπολογίες καταδεικνύουν ότι για πολλά σημαντικά θέματα, όπως το νέο Μητρό, για παράδειγμα, γεωγραφικών ενδείξεων, αποτελούν την καλύτερη προστασία σε ό,τι αφορά απάτη, σε ό,τι αφορά τη μετάφραση των γεωγραφικών ενδείξεων για τη διαπίστωση της προέλευσης των προϊόντων και για κάποια α, τέτοια δικαιώματα. Μπορούμε λοιπόν από εκεί να βρούμε καλές λύσεις και είμαι βέβαιη ότι και για εκκρεμή ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ευελιξία, την τροποποίηση των προσαρμοτημάτων, θα βρούμε κοινέ γραμμέ και συνένεση. Προσβλέπω λοιπόν πολύ στη συνεργασία. Μια παρατήρηση, επιτρέψτε μου κλείνοντα. Θα συζητήσουμε και στο μέλλον, θα πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά το βαθμό α, των, ε, των Αλλά δεν είναι εδώ το σωστό σημείο θα πρέπει να τα δούμε αυτά στα πλαίσια του κανονισμού για τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλα τα ενεπνεύματα. Σας ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω στις μελλοντικές μας συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Μπόιλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους και φυσικά την εισηγήτρια για το έργο της. Γνωρίζουμε ποιο είναι το σκεπτικό Τη ενημέρωση. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε την νομοθετική πρόταση με τη θήκη τη Λισαβόνα και να αρμονίσουμε τη διαδικασία ε, για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το πιο σημαντικό εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, προτείνει πιο ξεκάθαρες ρυθμίσει για την επισήμαση των αλκοολογών ποτών και εξαίρεση των στατικών ή διατροφικής για προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ πάνω από 2%. Θέλουμε τέτοια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε λήψη νομοθετικής πρότασης έχουμε καταθέσει τροπολογία στην έκθεση Αγιούζο για να, προλάβουμε, ε, για να περιλάβουμε τη δήλωση συστατικών και θρεπτικής αξίας. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Προς το παρόν ε, υπάρχει κενό και δεν γνωρίζουμε τις πληροφορίες παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει βάσιμους ε, λόγους για την έλλειψη αυτή, για την ε, παράληψη αυτή. Επίσης, ποιο είναι το μέγιστο όριο περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση ε, υπερβολικής ζάχαρης προς το τέλος της διαδικασίας παραγωγής προκειμένου να καλυφθούν κάποια ελαττώματα ορισμένων νεοπνευματοδών ποτών. προς όφελος των καταναλωτών είναι σημαντικό να έχουμε ακριβείς ε, επισημάνσεις, ακριβείς ετικέτες προϊόντων. Επίσης, ε, το ηλεκτρονικό μητρό αντικαθιστά πια το παράρτημα 3. Αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί και έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία. Θα πρέπει το νέο ηλεκτρονικό μητρό να έχει νομικό καθεστώς, να περιλαμβάνει όλα τα ε, προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων και να είναι συνεχώς προσβάσιμο. Επίσης το Μητρό θα πρέπει να εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε όλα ε, τα χαρακτηριστικά των ε, προϊόντων που έχουν ε, καταχωρηθεί με γεωγραφικές ενδείξεις και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνέπεια με τους τεχνικούς ε, φακέλους. Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερο από μία ονομασίες, ε, διαφορετική ορθογραφία, όπως το ελλαδικό Πούτσιν, ε, θα πρέπει να προσέξουμε τα θέματα της ορθογραφίας στις ονομασίες. Επίσης, τον τόπο Παρασκευής, γιατί μερικές φορές τα ενοπνευματόδη συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο, οπότε Μερικέ φορέ ο τόπο ε, θα πρέπει να τύχει εσεί, γιατί αυτό ευθύνεται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έχει μακροχρόνια ε, παράδοση. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σα ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο και οδηγητή στην αίθουσα. Περνάμε στους λοιπούς ομιλητές. Η κυρία Τελέ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το σύστημα προστασίας γεωργικών ενδείξεων είναι σημαντικό διακύβευμα της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των αχεγγύων ποιότητα, μα επιτρέπει να επανισορροπήσουμε τη θέση τη γεωργία στι εμπορικέ διαπραγματεύσει. Είναι σημαντικό το κείμενο των γεωγραφικών ενδείξεων, παρόλο που κάποια στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάσουμε πιο διεξοδικά. Το θέμα των υνοπνευματοδών ε, ποτών έχει κέρια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλο βάρος στις εξαγωγές μας. Ο προηγούμενος κανονισμός, το 110 του 2008, είναι ο τελευταίος γεωργικός κανονισμός που εναρμονίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και έγινε δεκτός από τους επαγγελματίες και η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξυγχρονίζει το κείμενο, πολύ ωραία, αλλά μέσω καταξιδότηση πράξεων αναλαμβάνει νέε αρμοδιότητε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβάλλει δύο πολύ σημαντικέ ε, τροποποιήσεις. Καταρχήν, καταργεί το παράρτημα 3 με τον κατάλογο των γεωργικών ε, ε, γεωγραφικών ενδείξεων και το αντικαθιστά από ένα ηλεκτρονικό online μητρό. Γιατί ε, όμως θα πρέπει να είναι λιγότερο αόριστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Μητρό και να μην έχει το δικαίωμα να το τροποποιεί μόνο με εκτελεστική πράξη. Επίσης, απαγορεύεται η μετάφραση των γεωγραφικών ενδείξεων στην ε, γλώσσα των χωρών που δεν έχουν το ίδιο αλφάβητο με μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει τη μετάφραση μόνο μέσω κατεξοδότηση πράξη, ενώ στο προηγούμενο κανονισμό προβλεπόταν συστηματική μετάφραση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιοριστεί απλώ στον εξυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του κειμένου και όχι στην ριζική τροποποίησή του με νέε διατάξει ε, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Και αυτή τη λογική ακολουθήσαμε και στην Επιτροπή Γεωργίας, όπου ήμουν η συγγήτρια της γνωμοδότησης. Είχαμε και την ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα το κείμενό μου υπερψηφίστηκε με μεγάλη ε, πλειοψηφία. Είχαμε σχεδόν ομοφωνία θα έλεγα, μία ψήφα μόνο κατά. Οπότε παρακαλώ τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος να, λάβει, να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Επιτροπής Γεωργίας, γιατί επαναλαμβάνω πρόκειται για ένα κανονισμό που αφορά την ετικετοθεσία, την επισήμαση, ένα τεχνικό κανονισμό για τα εινοπνευματόδηποτα και όχι ε, για ένα κανονισμό για την υγεία και προστασία των καταναλωτών ή ένα κανονισμό που αφορά τους κινδύνους από την υπερβολική ε, χρήση, την κατάχρηση αλκοόλ. Προσοχή λοιπόν να μην συγχαίουμε τα δύο θέματα. Ευχαριστώ την κυρία Πιλάρα Γιούζο, με την οποία είχαμε αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο ε, γραφείων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανα και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε και η συνάδελφος πριν από λίγο εδώ στο τέλος. Δεν είναι δυνατόν να κατατίθενται τόσες τροπολογίες που δεν έχουν να κάνουν τίποτα στη τελική ανάλυση με αυτή την τεχνική ρύθμιση που αποτελεί το αντικείμενο του κανονισμού. Δεν είναι ε, δυνατόν να χώνουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις ε, λίστες, στους καταλόγους, ε, τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν ταιριάζουν, δεν έχουν θέση εδώ στον κανονισμό. Πρόκειται για μια συζήτηση την οποία κάναμε και χθε ε, στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν ε, σχετικά νομοθετήματα τα οποία προετοιμάζουμε. Μάλλον σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει μια αυτορύθμιση. Θα τα ελέγξουν αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα έχουμε και την πρόταση πλευρά του κλάδου για το πώ και κατά να επαρκούν όλα αυτά. Κατά τα άλλα θα, ή τα άλλα θα προταθεί νομοθετική πράξη. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα, τον κανονισμό για τα ανεπνευματόδη, δεν έχουν θέση σε καμία περίπτωση αυτέ οι τροπολογίε. Γι' αυτό λοιπόν να τι απορρίψουμε, σα παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν να μπλέκουμε άσχετα μεταξύ του πράγματα. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες μας, ε, οι μου και να υποστρεφθούν... να βρούμε έναν όρο για τις ενώσεις, γιατί πιστεύω ότι δεν ε, ορίζονται επαρκώς ε, σε ό,τι αφορά επίσης το εθιλικό αλκοόλ. Είναι ο πνεύμα το οποίο αναφέρεται, θα πρέπει να μπορεί να είναι από γερική προέλευση, γιατί αναφέρεται ότι είναι από μπύρα, γιατί η μπύρα δεν είναι δεδομένο ότι αποτελεί γεωργικό προϊόν, παρότι είναι φυσικά, αλλά είναι και μεταποιημένο προϊόν με πολύ α, ενόπνευμα και θα μπορεί να μπορεί να συνεχιστεί αυτό το συγκεκριμένο εθελικό αλκοόλ για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τώρα την, τον, την περιεκτικότητα σε ζάχαρη των ενοπνευματοδών, είναι εργασία και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά τα άλλα θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα σε ό,τι αφορά την ε, χρήση ζάχαρης, αλλά να μην γίνεται στη τελευταία φάση αυτή και τέλος τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία διαθέτουμε και, διαθέτουμε και έχουμε πολλά τέτοια στο γερμανόφωνο κόσμο. Θα πρέπει φυσικά να μπορούμε να τα διατηρήσουμε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το Obst Brand, το Obst Layer για το πώς γράφεται το Likert για παράδειγμα Στη Γερμανία χρησιμοποιούμε τη γαλλική ορθογραφία. που Πρόκειται για παραδοσιακούς όρους και θα θέλαμε να διατηρηθούν και να υποστηριχθούν και σχετικές λοιπόν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Τώρα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ακούσουμε την κυρία Λουκατσόφνη. Από τη Γερική Διεύθυνση Αγγρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και την ε, κυρία Γιούζο, την εισηγητρία και την κυρία Ντελαέ από την Επιτροπή Άγκρη και τους ε, σκιώδες εισηγητές που συνέβαλαν όλοι στην εργασία για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζουμε τις τροπολογίες, τις πιο πολλές τροπολογίες και οι πιο πολλές εξ αυτών ε, ακολουθούν τον ίδιο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση στον τομέα των ίνοπνευματοδών που στο παρελθόν έδωσε ε, σημαντική όθηση στον κλάδο και συνέβαλε και στη συνολική ε, εικόνα του γεωργικού κλάδου σε ό,τι αφορά και τι γεωγραφικέ ενδείξει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί κατά τη σε ό,τι αφορά την πρόταση διάφορων ε, βουλευτών να καταργηθούν κάποιες από τις αρμοδιότητες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο των πνευματοδών. ποτών που υπόκειται στον κανονισμό. Ανησυχούμε για την δυνατότητα προσαρμογής των τεχνικών ε, διατάξεων όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη για σκοπό εξαγωγών. Και να αναφερθώ εδώ στο άρθρο 15, 5 και 16 της πρότασης. Αν καταργηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, ο κανονισμός θα καταστεί εντελώς άκαμπτος. Όπως ξέρετε, οποιαδήποτε καινοτομία δεν θα μπορεί να ενταχθεί στον κανονισμό. Με έναν τέλο πάντων αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο, όπως προαπαιτείται. Άρα, θα θέλαμε τουλάχιστον οι δυνατότητες κατηγοριοποίησης των ιονοπνευματικών ποτών και τεχνικών προδιαγραφών για την εξαγωγή να διατηρηθούν. Και να σας υπενθυμίσω από το 2008 και μετά κατά εξαίρεση του 110 του 2008 έχουν εγκριθεί 5 έως 10 τροπολογίες σε ό,τι αφορά την κατηγοροποίηση των ίνων πνευματοδών ποτών και για να εισαχθεί και μια νέα κατηγορία όπως είχε προταθεί από τις Ισπανικές Αρχές και τους Ισπανούς Παραγωγούς. Σε σε ό,τι αφορά το Πατσαράν. Να πω επίσης ότι συμφωνώ με όσους υποστηρίξαν ότι οι διτάξει που αφορούν τις ετικέτες σε ό,τι αφορά τα υλικά, τα συστατικά και την τρεπτική ε, αξία δεν ε, έχουν να κάνουν με το σωστό νομικό πλαίσιο. Όπως ακούσαμε ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια έκθεση για τα θέματα αυτά. Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους και έδωσε στον κλάδο ένα χρόνο να προσαρμοστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει λοιπόν την ρυθμιστική αυτή διαδικασία, θα εξετάσει κατά πόσο είναι επαρκής ή όχι και θα εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής μελέτης αντικτύπου. Και οι κανόνες αυτοί λοιπόν δεν ταιριάζουν στον κανονισμό αυτό. Δεν έχουν θέση εδώ παρά το γεγονός ότι ρυθμίζονται κάποιες πτυχές του καταλόγου των συστατικών που περιλαμβάνονται. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μπουν όλα σε ένα γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της, ε, του, της εθελικής ε, στη χρήση της ε, στην γεωργία, γεωργικής προέλευσης. Για να υπάρξει λοιπόν η σύνδεση μεταξύ του τομέα αυτού και της γεωργίας. Ε, για τα γεωργικά προϊόντα, δηλαδή που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1. Η πύρα δεν αποτελεί προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. Πρόκειται για μεταποιημένο προϊόν και ως ε, μεταποιημένο προϊόν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εθνική αλκοόλη για την ε, α, σε ό,τι αφορά την παραγωγή των προϊόντων. Δεν είναι θετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση εθελικής αλκόλη από μπύρα για την παραγωγή ενοπνευματοδών ποτών, γιατί θεωρώ ότι θα διακύβευε τα ενοπνευματόδη ποτά για την παραγωγή αυτών. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει πρόταση προς το Συμβούλιο για να, να επιτρέπεται η χρήση τη εθελικής αλκόλη ε, από μπύρας για άλλα αλκοόλουχα ποτά. Και εδώ πέρα αυτό οδηγεί και σε περαιτέρω σκέψη, σε κατατέθηκαν και σχετικέ τροπολογίε που περιορίζουν τη χρήση των κανόνων. Περιορίζουν μάλλον τους κανόνες για τη χρήση εθελικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης μόνο σε νυνοπνευματόδη. Και άλλα αλκοολούχα, όπως είναι τα αλκοπόψη, για παράδειγμα. αν καταργηθεί η διαταξή αυτή, δεν θα υπάρχει τέτοια διαταξή για τα ενοπνεύματα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και συμφετικό αλκοόλ. Θα ήταν λοιπόν μια πρόταση να περιοριστεί η χρήση αλκοόλ από μπύρα για άλλα αλκοόλουχα ποσά. Σε ό,τι αφορά το θέμα του αρθρού 13, το θέμα της μετάφρασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κατά του να επιτραπεί να προσθεθεί μετάφραση στις ετικέτες για σκοπούς εξαγωγής και προς την κατεύθυνση αυτή ε, έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιες εξουσίες και θέλουμε να ενταχθούν αυτά σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαστε κατά της ε, διάταξης ε, στην βασική πράξη κατευθείαν. Ωστόσο, να συστήσω προσοχή. Η μετάφραση κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων ήδη επιτρέπεται σύμφωνα με τους οριζοντίους κανόνες για τον κανονισμό που έχει να κάνει με τις πληροφορίες που χορηγούνται ε, στους καταναλωτές των 1169 του 2011. Αυτό γενικώ πώς επιτρέπεται. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι η μεταφράση των ονομάτων σε πλάγια γράμματα που δεν μεταφράζονται ή η μετάφραση της γεωγραφικής ένδειξης τα ονόματα αυτά, οι επωνυμίες αυτές δεν επιτρέπεται να μεταφράζονται στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή μπορεί να επιτραπεί η προσθήκη της μετάφρασης των ε, τίτλων αυτών, των ονομάτων αυτών στην ετικέτα και θα ήθελα να συστήσω να επιτρέπεται η μετάφραση και σε γλώσσες που αποτελούν και επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το να υπάρχει διάταξη σε μετάφραση, για να επιτρέπεται μεταφράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα επέτρεπε για παράδειγμα τη μετάφραση στα Ισπανικά. Για να γίνονται εξαγωγές προς την Λατινική Αμερική. Όσον αφορά τώρα την προέλευση, άρθρο 12. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπάθησε να δημιουργήσει μια διασύνδεση με κανόνες που ήδη υφίστανται και που ήδη εφαρμόζονται. Οι κανόνες αυτοί αφορούν, περιλαμβάνονται μάλλον στον τελωνιακό ε, ενωσιακό κώδικα. Στον προηγούμενο κανονισμό ε, υπήρχε αναφορά στον τόπο παρασκευής που ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένο τότε, αλλά δεν είχε λογική εφαρμοσιμότητα. Δηλαδή γινόταν απλώς ο ορισμός, αλλά δεν υπήρχε αντίστοιχη διάταξη που να επιβάλλει τη χρήση. Τώρα, το πρόβλημα ε, όσον αφορά ε, την αλλαγή του ορισμού του σημείου ε, προέλευσης ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί θα υπάρχει διτή μεταχείριση. Ε, μία όσον αφορά τον ενωσιακό ελληνιακό κώδικα, μία όσον αφορά τα ε, ινοπνευματόδη. Αυτό είναι μια οσον αφορα τον ενωσιακο ελληνιακο κωδικα μια οσον αφορα τα εινοπνευματώδη. αυτο ειναι μια προειδοποιηση που σας κάνω. Μπορεί να συζητηθεί βέβαια, αλλά αναφέρομαι στο πρόβλημα αυτό, το οποίο, στο θέμα αυτό το οποίο ενδεχομένω θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Όσον αφορά τη γλύκανση. κυρίως ε, για τις ε, ε, κατηγορίες εμβολών 1 έως 14 του παραρτήματος 2. Καθαρά είναι πνεύματα. Η Κομισιόν μπορεί να συμφωνήσει με τον ορισμό μεγίστων όριων. Δεν το κάναμε γιατί αυτό είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Κάθε χώρα έχει δικιά της νομοθεσία όσον αφορά τα θέματα αυτά και ε, ο κανονισμός αυτός όμως θα πρέπει να ε, επιτύχει ένα ικανό επίπεδο εναρμόνισης ε, εντός των νομοθετικών διαταγμάτων και απαιτήσεων στα κράτη-μέλη. Μπορεί να υπάρχει ένα ε, μέγιστο αποδεκτό όριο χρήσης γλυκαντικών ουσιών, αλλά να είναι τέτοιο που να οδηγήσει σε ένα ε, νόμο που να μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πιο περιοριστικοί κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν σε εθνικές επικράτειες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάποιες ε, προσπάθειες απλούστευσης για τα μείγματα to eliminate geographical indications from the possibility to μείγματα και αναμίξεις Ε, θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο, αλλά θα έπρεπε να αλλάξουν ε, οι τρέχουσες ε, πρακτικές, γιατί υπάρχουν πολλά μείγματα τύπου Grand Marnier, ας πούμε. Το Grand γίνεται με κονιάκ, το οποίο είναι συγκεκριμένης προστατευμένης προέλευσης και επομένως θα βρισκόταν να είναι παράνομο. Ε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ε, κάποιες παρανοήσεις ε, όσον αφορά τα πλάγια γράμματα. Όταν ένα όρος στο παράρτημα 2 είναι στα πλάγια δεν σημαίνει ότι προστατεύεται ως τέτοιο, σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταφραστεί για να ε, ε, προστατευτεί ε, η αναφορά σε εθνικές ας πούμε παραγωγές, το λικέρ ή λίκουορ στα γερμανικά ή στα αγγλικά. Η καλύτερη λύση θα ήταν να γίνει αποδεκτή η χρήση του όρου λικέρ σε πλάγια γράμματα και λικέρ σε όρθια γράμματα, μη πλάγια, που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφραστεί. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το σημείο διμερό αν θέλετε. Ε, επίσης έχουμε και κάποιους προβληματισμούς ε, όσον αφορά μια γνώμη, ε, η οποία, μια γνωμοδότηση που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Γεωργίας σύμφωνα με τις τροπολογίες ε, μονάχα ένα ε, εινοπνευματόδες μπορεί να εμπέσει στην ε, κατηγορία αυτή των παραπομπών που υπάρχουν ήδη για τα εινοπνευματόδη. Έχουμε και ένα άλλο θέμα σχετικά με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας. Υπάρχει μια τροπολογία η οποία έχει υπερψηφιστεί που απαγορεύει ε, ε, ε, ε ψεύτικα πρόσθετα ουσίας για τα Ε, Εμείς απαγορεύουμε τα στοιχεία αυτά. Ας πούμε υπάρχουν κάποιες μπύρες ε, με ε, ουσίες ε, τότε εάν δεν πούμε ότι αυτές οι μπύρες είναι πραγματικά υνοπνευματόδη, τότε θα ανοίξουμε το δρόμο να χρησιμοποιηθούν μη φυσικές ουσίες γεύσης. Και επομένως σε όλα τα ποτά ε, σε όλα τα ποτά τα ενοπνευματόδη ε, θα πρέπει να είναι σαφές ότι ουσίες ενίσχυσης γεύσης θα πρέπει να είναι πραγματικές και όχι ψεύτικες. Ε, σε άλλα ποτά όταν γίνεται αναφορά σε flavor, σε γεύση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να γίνει ένα κέικ ας πούμε, όχι όμως είναι ο Μπορεί ε, να επιτραπεί η χρήση ε, ε, ψεύτικων επιγεύσεων μόνο σε άλλα είδη και όχι στα υνοπνευματόδη. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις θα μιλήσει ο συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όπως και η συνάδελφός μου Εγώ λέγομαι Λούκα Τσαμφώνη και ασχολούμαι μονάχα με το κεφάλαιο που αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Όσον αφορά λοιπόν τις γεωγραφικές ενδείξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετικά δέχεται πολλές από τις προτινόμενες τροπολογίες. Θα ήθελα άμεσα να πω ότι η Κομισιόν είναι υπέρ των τροπολογιών οι οποίες στόχο έχουν να διευρύνουν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των ακόμα και όσον αφορά ε, τις, ε, ε, τα, τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε διαμετακόμιση εντός, του, εντός της τελωνιακής επικρατείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία απέτηση η οποία είναι πάρα πολύ έντονη από τον τομέα ε, των υνοπνευματοδών. Επίσης, ε, υπάρχει ε, η προστασία αυτή όσον αφορά τα εμπορικά σήματα trademarks. Όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έφυξε η κυρία Αγιούσο δηλαδή να εξηγήσει αυτή τη διχοτομία ανάμεσα ε, ε καταχωρημένες και προστατευόμενες γεωργιακές προελεύσεις από το εξής. Ε, στον τομέα των spirit drinks, εμείς δεν έχουμε όπως στον τομέα άλλων γεωργικών προϊόντων ε, και όπως και στον τομέα του κρασιού, δύο διαφορετικές κατηγορίες, Προστατευόμενη και καταγεγραμμένη ονομασία προέλευσης. Προ, ε, προστατευμένη γεωγραφική προέλευση και ε, ε, προστατευμένη γεωγραφική περιοχή. στην περίπτωση της ένδειξης περιλαμβάνονται στην προκείμενη περίπτωση όλες οι προστασίες. Όταν έχουμε μία γεωγραφική ένδειξη. Όταν λέμε προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη και μιλάμε για γεωγραφική ένδειξη στα ε, ινοπνευματώδη, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το PGI, γιατί αυτό το ακρονίμιο αναφέρεται ε, στην, ε, στις προστατευόμενες ε, περιπτώσεις για τα τρόφιμα και για το κρασί. Ενώ εδώ εμείς θέλουμε να πούμε προστατευόμενο με την έννοια της περιγραφής της γεωγραφικής περιφέρειας που ακριβώς λέει ποια είναι η γεωγραφική ένδειξη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του τομέα έτσι ώστε να ε, ε, ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να μην μιλάμε για protected geographical indication για τα υνοπνευματόδη. Γιατί είναι προφανές ότι θα μπορούσε να προκύψει ε, μία σύγχυση με την ένδειξη PGI για τα τρόφιμα. Ε, επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε ε, protected με registered, προστατευόμενο με καταχωρημένο, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε, ε, σε παρεξηγήσεις, σε παρανοήσεις. Ίσως θα μπορούσε στο μέλλον να δημιουργηθεί το RGI, δηλαδή Registered Geographic Indication, καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη. Όμως, εμείς θεωρούμε ότι μέσω μιας μικρής τροποποίησης ε, του ε, ορισμού της γεωγραφικής ένδειξης μπορούσε να λυθεί το θέμα. Δηλαδή να πούμε ότι μιλάμε για γεωγραφικές ενδείξεις IG οι οποίες καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες και προστατεύονται κατά την έννοια των διατάξεων του λόγου ε, λόγω κανονισμού. Έτσι να νοείται δηλαδή κάθε φορά η γεωγραφική ένδειξη ε, για τα εινοπνευματόδη. Επομένως δεν θα υπάρχει λόγος να διαχωρίζουμε σε προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις και σε καταχωρισμένες ε, ενδείξεις. Ε, θα ξέρουμε ότι πρόκειται για γεωγραφική ένδειξη η οποία και είναι καταχωρισμένη και είναι προστατευμένη. Αλλαγή λοιπόν της διατύπωσης στους ορισμούς στην αρχή του κειμένου. Αυτό μπορούμε να το διευκρινίσουμε και περαιτέρω. Να επιστρέψω τώρα στις τροπολογίες. Υπάρχουν 46 τροπολογίες οι οποίες κατά τη δική μας άποψη ε, αντιτίθενται στην αρχική ιδέα της πρότασης. Ε, θα πω δύο λόγια λοιπόν για τις τροπολογίες αυτές. Και θα ξεχωρίσω τα προβλήματα σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες παρουσιάζουν διαθρωτικά νομικά προβλήματα ε, και που είναι ασύμβατες με την ισχύουσα νομοθεσία που είναι ασύμβατες επίσης και με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο και που ε, ε, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το πεδίο εφαρμογής όλης της πρότασης. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες οι οποίες είναι επίσης ε, σημαντικές ε, και προβληματίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ας πούμε μειώνουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια του συστήματος ε, ή δυσχεραίνουν τη διαχείριση του συστήματος αλλά αυτές είναι λιγότερο σοβαρές κατά κάποιο τρόπο τροπολογίες. Έχουμε ας πούμε την τροπολογία 176 που συνδέεται και με την τροπολογία 315 όπου προτείνεται να διαγραφεί η λέξη reputation όσον αφήμη, όσον αφορά τη γεωγραφική ένδειξη. Η Κομισιόν θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι μια τέτοια τροποποίηση αντιτίθεται στην συμφωνία TRIPS, ε, τις απαιτήσεις TRIPS ε, του διεθνούς, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εμπορίου. Θα αντιτίθεται λοιπόν σε αυτήν την συμφωνία ε, τρίψε που, απαιτεί, ε, που αποτελεί συγγνώμη, τη βάση για, την, ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα γιατί αυτό ισχύει και για όλους τους τομείς και για, το, για τα τρόφιμα και για το κρασί και για τα υνοπνευματόδη και ακριβώς θα αντιτίθεται σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες και θα διακινδυνεύαμε στο μέλλον να διαγραφούν στο μέλλον γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες βασίζονται παραδοσιακά και μόνο στην φήμη στη γνώση του προϊόντος. Επομένως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έχουμε μια άλλη τροπολογία, τροπολογία υπαριθμών 14. όπου το αίτημα από τρίτη χώρα ε, να λαμβάνεται υπόψη μονάχα από τις ε, τοπικές αρχές. Δηλαδή, οι ε, παραγωγοί των τρίτων χωρών δεν θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν άμεσα στην Κομισιόν το αίτημα. Υπάρχει αυτή η διάταξη ήδη στον κανονισμό για τα γεωργικά προϊόντα και Αποτέλεσε αντικείμενο διαδικασίας εντός του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορίου ε, έτσι ώστε ε, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν να μην μπορέσουν να αποτελέσουν δεσπόζουσα δύναμη η οποία θα μπορούσε να πιέσει τις αρχές έτσι ώστε να απαγορεύσουν στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες να στείλουν το αίτημα άμεσα και να μην περάσουν οπωσδήποτε ε, από ε, κάποια κρατική αρχή. Υπάρχει και μια άλλη τροπολογία η οποία αντιτίθεται στον τρόπο λειτουργίας. Είναι η 338 και αφορά το άρθρο για τις ε, προσφυγές και τις αντιθέσεις. Εκεί ε, γίνεται λόγος ε, για ε, ένα απλό, για μια απλή ταχυδρομική αποστολή, αλλά εδώ εμείς δεν παίρνουμε σαν αναφορά αυτό, εμείς λαμβάνουμε υπόψη είτε την ημερομηνία της αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε την ημερομηνία που καταγράφεται στο τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία. Για το κρασί, ας πούμε, έχουμε την εφαρμογή που οποία λειτουργεί. Επίσης υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες θέλουν να δώσουν στην Κομισιόν ε, εξουσία για ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξης, αλλά για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είναι ας πούμε έγκριση κατ ε, ε, έγκριση για ένα νέο κανονισμό για ένα νέο όνομα ή για διαγραφή παλαιού συστήματος. Αυτές είναι νομοθετικές πράξεις συγκεκριμένες και θεωρούν και η Κομισιόν θεωρεί ότι η εκτελεστική πράξη είναι η πρεσίκουσα νομική μορφή. Όσον αφορά την, ε, την τήρηση αρχείου ε, διατήρηση με την έννοια της επικαιροποίηση ε, του αρχείου και επομένως ε, είτε να διαγραφούν παλές ονομασίες είτε να προσθεθούν νέες. Επίσης υπάρχει και μια τροπολογία η οποία είναι πολύ σημαντική. είναι η τροπολογία η οποία αφορά την δυνατότητα κατηχώρησης ομονίμων. Ε, δηλαδή ε, ομώνυμα σε σχέση με ονόματα, ονομασίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί. Ε, υπάρχει η διάταξη TRIPS 130 που λέει ότι μία ομώνυμη ονομαθεσία που μπορεί ήδη καταχωρημένη, η οποία μπορεί να δημιουργήσει παρανόηση στο πνεύμα των καταναλωτών δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η τροπολογία 359 ε, ε, θέλει να επιτραπεί η καταχώρηση. Αυτό όμως ε, μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί μελλοντικά να έχουμε καταγεγραμμένη μία ριόχα από την Αργεντινή ή μία σαμπάνια από τον Καναδά. Πρόεδρο. Λυπούμε. παρακαλώ βάλτε κάπου τελεία γιατί έχει προχωρήσει η ώρα. Thank you. Okay, thank you. I will, try to summarize. Yeah. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να τα πω σύντομα. Υπάρχει άλλη μια σημαντική τροπολογία η οποία θέλει, ε, ζητά κατάργηση των ε, ε, σωμάτων ελέγχου, control bodies, οργανισμούς ελέγχου όσον αφορά δηλαδή τον έλεγχο της συμμόρφωσης, ε, ε, όσον αφορά ε, το... όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Ε, και εδώ αναφερόμαστε σε τρίτες χώρες και επομένως αντιτίθεται ε, στις ε, αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ήδη στο πάνελ υψηλού επίπεδου και όπου καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τρίτων χωρών. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η τροπολογία 321 γιατί αρνείται στην Κομισιόν την δυνατότητα να εγκρίνει τις διαδικασίες για τις τροποποιήσεις. Είναι διαδικαστικά βεβαίως τα στοιχεία αυτά αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί αυτή η πρόταση της Κομισιόν καθορίζει βάση της ε, επικουρικότητας ε, την ε, δυνατότητα εξουσιοδότησης στα κράτη-μέλη πολλών αρχών διοικητικών. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες οι οποίες επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα, τα αναφέρω εντάχει. Υπάρχει η τροπολογία ας πούμε η οποία μειώνει τον ε, χρόνο ε, ελέγχου εξέτασης ε, της Κομισιόν από 12 σε 6 μήνες. Η Κομισιόν επιμένει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την εξέταση των ετοιμάτων, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν η Κομισιόν υποχρεωθεί να περιοριστεί στους 6 μήνες τότε η Κομισιόν ζητάει ε, η ανάλυση που υποχρεούται η Κομισιόν να κάνει να είναι λιγότερο ε, ε, σε βάθος και λιγότερο λεπτομερής από αυτή που προβλήπεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή να περιοριστεί, να, να, να, μην υπάρχει έλεγχος πέραν του ελέγχου περί προδήλου σφάλματος. Επίσης ε, η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι γενικά μπορεί να είναι θετικό κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης ε, και στο αρχείο αλλά και στο Μητρό και στις διεθνείς συμφωνίες αλλά δεν έχουμε χρόνο και επομένως δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, με μακρηγορήσατε αρκετά σήμερα. Μιλήσατε πολύ περισσότερο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ότι ευρωβουλευτές. Και πάλι ο λόγος στην εισηγητριά μας την κυρία Γιούσο για τα τελικά σχόλια της σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι λακωνική γιατί ε, χαίρομαι που είχε το χρόνο να μιλήσει εκτενώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλωστε είχα κάνει και εγώ ερωτήσεις. Ευχαριστώ θερμά τους και όδη την κυρία Τελαέ, την εισηγήτρια της γνωμοδότης Επιτροπής Γεωργίας, δυστυχώς έφυγε. Σημείωσα σχολαστικά όλα τα σχόλια που ακούσαμε και τις παρατηρήσεις και θα συνεχίσω τις επαφές με τους και ηγητές την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να εκπονήσουμε συμβαστικές τροπολογίες και να τις στείλουμε στους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιούσο, εμείς ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 28 Νοεμβρίου και έτσι διεκπαιρεώσαμε την πρωινή μας ε, συζήτηση, συνεδρίαση. 23 Οκτωβρίου στο Στρασβούρο θα είναι η επόμενή μας συνεδρίαση, μια και δεν υπάρχουν διάφορα. Και 6 Νοεμβρίου η επόμενή μας συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Καλό σας μεσημέρι.